Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Αλίας. Καταρχήν η διάταξη. Υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις που θα σας προτείνω. Είναι δύσκολο να καταρτήσει κανείς την ημερήσια διάταξη αυτήν την ε, αυτής της Επιτροπής, γιατί υπάρχουν πολλές αιτήσει για αλλαγέ. Και ξέρω ότι πολλοί βουλευτές ε, έχουν και άλλες συνεδριάσεις τις οποίες πρέπει να παραστούν και πολλές φορές αλλάζουν την ε, σειρά εμφάνισή τους ή τουλάχιστον ζητούν να αλλάξουν τη σειρά εμφάνισή τους. Λοιπόν, έχουμε τα εξή ε, να σας αναφέρω. Το σημείο 15 που θα ήταν η επίσκεψη του κυρίου Άσφιλτ από τον Καναδά έχει ακυρωθεί. Το θέμα αυτό λοιπόν δεν θα το αντιμετωπίσουμε. Και έτσι το, επίσης το σημείο 9 του κυρίου Ρωμέβα για την τροποποίηση του κανονισμού 302-209 για τον ε, ερυθρό τόνο που κανονικά θα το, βλέπαμε, θα το αντιμετώπιζαμε σήμερα θα πάει στη θέση του σημείου 15 στη θέση του Καναδού Υπουργού. Έχουμε όμως προσθέσει ένα σημείο 9α του κυρίου Μπεσέτ στη σημερινή ημερήσια διαταξή και επίσης για τις ψηφοφορίες που προβλεπόταν να γίνουν αύριο στις 9 θα γίνουν στην πραγματικότητα στις 11 αύριο το πρωί η ψηφοφορία αντί για 9. Υπάρχουν αντίρρησεις για τις τροποποιήσεις αυτές. Ωραία. Θεωρείτε ότι έχει εγκριθεί η ημερησία διάταξη με αυτές τις τροποποιήσεις. Πρακτικά. 20-22 Μαρτίου, ως ήθιστε, εάν μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάρξει καμιά αντίρρηση, θα θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί. Ανακοινώσει του Προέδρου, μηδέν. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Περνάμε κατευθείαν στο σημείο υπαριθμών 4, τροποποίηση του κανονισμού 1967-2006 του Συμβουλίου σε σχέση με τα μέτρα διαχείρισης για την αηφόρο εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο. Στις 10 Οκτωβρίου έκανε μια παρουσίαση για το θέμα αυτό η Κομισιόν. 19 Δεκεμβρίου είχαμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό το Δεκέμβριο και τώρα η κυρία Ρόσπαχ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της και της δίνω αμέσως το λόγο. Κυρία Ρόσπαχ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για την ευθυγράμμιση ενός κανονισμού που ήδη έχει κατεθεί και είναι υποσυζήτηση εδώ και κάποιο καιρό και είναι, πρόκειται απλά για την ευθυγράμμιση με τη διαδικασία της Λισαβόνας. Βιώσιμη για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων στη Μεσόγειο θάλασσα ε, να τρέχει στο 2003, οπότε έγινε η πρώτη αλλαγή του κανονισμού για να, σε σχέση με τον πρώτο κανονισμό που είχε εκδοθεί το 1994. Εγκρίθηκε λοιπόν ο λόγω κανονισμός μόνο το 2006. Λόγω των ε, γεωλογικών χαρακτηριστικών είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς το ότι η Μεσόγειο θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα πράγμα που σημαίνει μέτρα συντήρησης και όχι μόνο μπορικά μέτρα. Τώρα, η πίεση από την αλίευση στην Μεσόγειο σημαίνει πως διάφορα είδη είναι υπό απειλή εξαφάνισης. Οι επιστήμονες ε, δείχνουν, ε, μάλλον έχουν υποδείξει κάποια είδη, ενώ κάποια άλλα είδη δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί. Δηλαδή δεν έχουμε καμιά ιδέα για το ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων, των αληφτικών αποθεμάτων. Μόνο η έρευνα που έχει γίνει είναι σχετικά με τον τόνο και η παράνομη αλληλεία τόνου είναι μια πηγή ανησυχίας. Όταν υιοθετήθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας, εισήχθη ένα νέο σύστημα για όλα τα θεσμικά όργανα και χρειαζόταν ευθυγράμμιση της, ε, των σχετικών νομοθετικών κειμένων. Και αυτή είναι η πρώτη πρόταση για τον τομέα της αλληλείας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η ευθυγράμμιση. Το Ευρωκοινοβούλιο τοποθετείται επί ίσης ώρες με το Συμβούλιο για τις περισ... είναι ισότιμοι συνομοθέτες για τις περισσότερες νομοθετικές διατάξεις και υπάρχει έτσι μια νέα ιεράρχηση κανόνων. Η πρώτη, το πρώτο στάδιο είναι η τακτική νομοθετική διαδικασία, όπου όπως σας είπα είμαστε επίση ώρες με το Συμβούλιο. Το δεύτερο επίπεδο είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης προς την Κομισιόν, ώστε να μπορεί να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής. Αυτές τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις τις γνωρίζετε πλέον όλοι. Και αυτό είναι έργο της Κομισιόν. Τώρα έχουμε και το τρίτο επίπεδο που είναι οι πράξεις εφαρμοστικέ. Από τη στιγμή που ισχύουν οι ίδιοι όροι και συνθήκε σε όλε τι χώρε Εδώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απλά έχουν το δικαίωμα παρατήρηση τη υιοθέτηση αυτών των κειμένων, των πράξεων των εφαρμοστικών. Το Κοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο δεν αποτελούν μέρο αυτή τη διαδικασία. Πρέπει αυτό λοιπόν να το γνωρίζουμε και να το προσέξουμε. Δύο διαφορετικές πράξεις λοιπόν, η κατεξουσιοδότηση και οι εφαρμοστικές. Η Κομισιόν όμως έχει ευθυγραμμίσει μόνο κάποιες ρήτρε του κανονισμού, αυτές δηλαδή που υπήρχαν στον παλιό κανονισμό, αναφέρονταν στην παλιά διαδικασία επιτροπολογίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνεται υπόψη επίσης όρις όπως το Συμβούλιο, όπως δηλώνει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό γιατί η ευθυγράμμιση δεν αλλάζει το περιεχόμενο της ε, ε, νομοθεσίας. Μόνο η νομική πράξη που θα επιλέξουμε. Στην έκθεσή μου και στη συζήτηση με τους Κεώδης και τις ε, νομοθετικές υπηρεσίες συμφωνήσαμε με την Κομισιόν, συμφωνούμε μάλλον με την Κομισιόν και στη συγκεκριμένη έκθεση εξετάζουμε την 8η πρόταση και εγώ έχω κάνει κάποιες τροπολογίες, 27 συγκεκριμένα. Θα σας πω ποιες είναι οι πιο σημαντικές. Ορισμένοι μπορεί να πιστεύετε ότι δεν είναι κέρυες, αλλά κατά τη γνώμη μου Αξίζει να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή μας. Γιατί εδώ έχουμε μια δυνατότητα να εισάγουμε μέτρα συντήρησης και την βιωσιμότητα στον τίτλο. Και θα ήθελα οι συνάδελφοι να στηρίξουν αυτή την πρόταση, να μπουν δηλαδή στον τίτλο αυτές οι λέξεις. Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων. Γιατί η νομοθεσία περί δεν ε, θα πρέπει μόνο να ορίζει τον τρόπο εκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων, αλλά και τη διατήρηση ε, και τη βιώσιμη εκμετάλλευση αυτών. Επίσης, στα παραρτήματα ε, θα πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με την Κομισιόν που θέλει να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμοστικές πράξεις για τα παρατήματα, γιατί τα παρατήματα είναι αναπόσπαστο τμήμα της, νομοθε... της νομοθεσίας. Στην έκθεσή μου λοιπόν προτείνω να αλλάξουμε την πρόταση της Κομισιόν έτσι ώστε τα παρατήματα να αποτελούν τμήμα της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμμετέχουν. Ε, πρόκειται για τις τροπολογίες 10, 11 και 12. Οι εφαρμοστικές πράξεις επίσης θα πρέπει να είναι περιορισμένου χρόνου. Αυτή τη στιγμή είναι άνευ χρονικών ορίων, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μην μπορούν να τις επηρεάσουν. Γι' αυτό και προτείνω μια τριετή περίοδο που να μπορεί να παραταθεί Στην πρόταση της Κομισιόν υπάρχει λοιπόν ευθυγράμμιση 8 ε, ρητρών. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να ευθυγραμμίσει πλήρως την πρόταση για όλες τις ρήτρες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δίνουν μόνο στο Συμβούλιο το δικαίωμα να αποφασίζει, πράγμα το οποίο δεν είναι πλέον δυνατόν υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στις περισσότερες λοιπόν περιπτώσεις προτείνω να χρησιμοποιηθεί το μέσο της κατεξουσιοδότηση ε, πράξεως, αλλά στις περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη θέλουν να εισάγουν εθνικού επίπεδου μέτρα που θα ελέγχονται από την Κομισιόν, προτείνω εκεί η Κομισιόν να μπορεί να λειτουργήσει με κατεξουδότηση πράξης, καθώς και στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη θεωρούνται ανεπαρκή. Όταν μιλάμε για τα κράτη-μέλη και για νέους περιοχές όπου δεν θα πρέπει να γίνεται αλληλεία ΕΕ. εκεί που συμμετέχουν και γειτονικέ χώρες. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εμπλέκεται στη διαδικασία και η διαδικασία αυτή να είναι τμήμα της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Υπάρχουν και κάποια χρονικά όρια. τα οποία έχουν ήδη εκπνεύσει και νομίζω πως αν παραταθούν τα χρονικά όρια θα γίνει συζήτηση που δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της νομοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, δεν πιστεύω πως θα ήταν σκόπιμο να καταργηθούν τα χρονικά όρια. Άρθρο 14, παράγραφος 3 μπορεί να ερμηνευθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Συμβούλιο να μπορεί να παρατείνει τα χρονικά όρια της προθεσμίας. Γι' αυτό και προτείνω να διαγραφεί αυτό το χρονικό όριο που ήταν το 2010. Και τέλος, σύντομα, να σας πω πως ε, όντως η, η Μεσόγειος είναι ιδιαίτερη θάλασσα και αυτό θα πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη γύρω από την Μεσόγειο να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή της νομοθεσίας, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει καθόλου μέχρι τώρα. Πιστεύω, ελπίζω ότι η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα αποτελέσει μεταρρύθμιση και για τη Μεσόγειο, ώστε να έχουμε πλέον βιώσιμη αλληλεία στην Μεσόγειο και νομοθεσία που θα γίνει δεκτή και θα εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη και τους αλληλείς τους στην Μεσόγειο. Και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος λέει. Κυρία Φράγα, έχετε το λόγο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σιγητρή γιατί έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά σε αυτό το θέμα το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα κάπως βαρετό θέμα γιατί η προσαρμογή στην επιτροπολογία δεν είναι ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Νομίζω ότι η συγγήτρια έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία και με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε μια πλήρη προσαρμογή και όχι απλώς μια εν μέρη προσαρμογή όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν για την εκχώρηση εξουσιών νομίζω το Κοινοβούλιο έκανε μια σωστή επιλογή για τα σημεία που πρέπει να παραμείνουν στη συναπόφαση και αυτά που πρέπει να είναι εξουσιοδότηση πράξης. Όλα τα παρατήματα με τις λεπτομέρειες και τα ειδικά μέτρα, αυτά είναι θέματα τα εγώ θα προτιμούσα να μείνουν στον τομέα της συναπόφασης και όχι κατεχώρηση όπως λέει η συγγήτρια. Αλλά είναι πολλά θέματα τα οποία είναι περίπου θέματα τύπου και όχι θέματα ουσίας, όπως είναι η τροποποίηση του τίτλου. Αν θέλουμε να αλλάξουμε βέβαια τον τίτλο του νομοθετήματος, εφόσον κάνουμε μονάχα μια διαδικασία επιτροπολογίας, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, γιατί δεν είναι ο στόχος αυτού του εγχειρήματο. Όταν τώρα στο μέλλον αλλάξουμε εκβάθρον ή τροποποιήσουμε τα βασικά στοιχεία του κανονισμού, τότε μπορούμε να αλλάξουμε και τον τίτλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα τύπου και όχι ουσία. Εγώ δεν θα ήθελα όμω τώρα να γίνει αυτή η μετατροπή του τίτλου. Κατά τα άλλα είναι θαυμάσια η εργασία της κυρίας Ρόσπαχ. Εμείς ως πολιτική ομάδα θα ακολουθήσουμε την, τον δρόμο που χάραξε η κυρία Ρόσπαχ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Κυρία Ρόσπαχ θέλετε να επανέλθετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να μπορώ να έχω την υποστήριξη των συναδέλφων μου. Κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ προκειμένου να συντάξω μια έκθεση η οποία θα αναποδεχθεί από όλου και θέλω να έχω ένα πολύ καλό διάλογο με την κυρία Φράγκα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε σίγουρα τη μεταρρύθμιση του κανονισμού αυτού. Τι θα κάνουμε όμως το ενδιάμεσο διάστημα, αυτό είναι το ερώτημα που σας θέτω. Υπάρχουν και άλλοι θαλάσσιοι πόροι πέρα από τους ελευτικούς με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συνένεση και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι μέχρι τι 7 Μαου το μεσημέρι. Επόμενο σημείο, σημείο 5, ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Διακόπτεται ο πρόεδρο. Α, δεν είχα δώσει το λόγο στην Κομισιόν. Πώ θέλει να μιλήσει η Κομισιόν. Θέλετε να παρέμβετε, κύριε τα ε, The ε, Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη μέση διάταξη και δεν νομίζω ότι οι αρμόδιοι συνάδελφοι για το θέμα αυτό είναι παρόντες. Σε αυτή την περίπτωση δεν άλλαξε η Μέση διάταξη, αυτό το σημείο έμεινε στη θέση του τώρα. Αν δεν είναι για άλλους λόγους οι αρμόδιοι, το καταλαβαίνω, αλλά εμείς δεν ευθέμε που αλλάξαμε την Μέση διάταξη. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν, σημείο 5, ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής αλληλευτικής συγγνώμη πολιτικής η παρουσίαση έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου. Ξέρετε ότι το έγγραφο εργασίας παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα, τον Ιανουάριο συγγνώμη, Έγινε πρώτα μια παρουσίαση τον Νοέμβριο και μετά το έγγραφο εργασία παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαβράκο για να μα παρουσιάσει την έκθεση, το έγγραφο εργασία του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και επειδή το θέμα ήδη έχει συζητηθεί εκτενώς όλους αυτούς τους μήνες από την Επιτροπή θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η ανακοίνωση της Επιτροπής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτάσεων και στο σχέδιο της έκθεσης που σας παρουσιάζεται σήμερα προσπάθησα να αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία. Πρώτο σημείο, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συμφωνώ με το στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως μέσο για τη σταδιακή εξάλληψη της υπεραλίευσης και την επίτευξη της αηφόρου διαχείρισης των αλλιευμάτων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην άμεση εφαρμογή του στόχου FMSY που κρίνεται πιο ρεαλιστικός και που σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα για την ανάκαμψη των αποθεμάτων. Ως προ το μέτρο αυτό τονίζονται οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη ως προς την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων και τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων καθώς και στην περίπτωση της μεικτή αλίας. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις της πολυειδούς αλίας και να παρέχει στα κράτη-μέλη επαρκή λιγοτεχνική και οικονομική υποστήριξη προς το σκοπό Τονίζεται η σημασία των ερευνητικών συνεργασιών Thank you. και τη συμμετοχή των αλλιέων σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο σημείο είναι η απαγόρευση των απορρίψεων. Ως προς την απαγόρευση των απορρίψεων αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα παύσης αυτής της πρακτικής καταρχήν ω πατάλη πόρων και ω πρακτικά επιζήμια για το οικοσύστημα, αλλά και για την ασφαλή διεξαγωγή ζωτική σημασία αξιολογήσεων. Προτεραιότητα ωστόσο οφείλει να είναι η ανάπτυξη, η ανάπτυξη επιλεκτικών μεθοδών αλληλείας, που θα μειώσουν τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα για όλους τους τύπους της αλληλείας. Καλείται η Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο να προωθήσει τις συνέργειες μεταξύ των επιστημόνων και των αλλιέων στην πράξη, η εφαρμογή αυτού του μέτρου χρειάζεται προσοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην μεταφέρουμε το πρόβλημα από τη θάλασσα στην ξηρά και έτσι καταλήξουμε από ανεπιθύμητα αλλιεύματα στη θάλασσα να έχουμε ανεπιθύμητα αλλιεύματα στη σταριά. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επίσης, καθώς η νέα αλλιευτική πολιτική που χαράζουμε θα εφαρμοστεί για τα επόμενα 10 χρόνια και οφείλουμε να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και ρεαλιστικά μέτρα που θα έχουν την μέγιστη δυνατή υποστήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται φρόνιμο να εκπονήσει η Επιτροπή πιλωτικά σχέδια ώστε να εντοπιστούν οι τεχνικές δυσκολίες και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά, εκφόρτωση και διαχείριση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων καθώς και να συνεκτιμηθεί το διοικητικό κόστος και οι δυσκολίες της επιθεώρησης της αλλιείας. Το μέτρο της εμπορίας των παρεμπιπτόντων αλλιευμάτων θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μην καταλήξουμε παραδόξως στη δημιουργία μιας παράλληλης αγοράς. Το τρίτο σημείο είναι οι μεταβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις. Ως προς το ζήτημα αυτό το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ των μεταβάσιμων παραχωρήσεων θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ως το μοναδικό μέτρο για τη μείωση της αλλιευτικής ικανότητας. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη μια αξιολόγηση της αλλιευτικής ικανότητας του στόλου για να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ακριβή κατάσταση της πλεονάζουσας αλλιευτικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα στοχευμένα μέτρα για τη μείωσή της. Οι ανησυχίες για συγκέντρωση και δημιουργία μονοπωλίων είναι έκδηλες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράκτια αλλία και την αλληλεία μικρής κλίμακος που αποτελούν τα πλέον απειλούμενα από οικονομική άποψη μέρη του κλάδου αλλά και εκείνα που παρέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας κατά την βασική οικονομική δραστηριότητα στις παράκτιες περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον σχεδιασμό ενός τέτοιου μέτρου παρέχοντας ρήτρες διασφάλισης και εχέγγυα για την προστασία της μικρής κλίμακος ελίας. Τέταρτον, οι υψηλές τιμές πετρελαίου. Από συζητήσεις μου με φορείς του κλάδου, οι υψηλές τιμές πετρελαίου αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους ελληνείς ειδικά αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που ο κλάδος της αλληλείας δοκιμάζεται. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου ώστε να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντολογικής και κοινοοικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου και ίσως θα πρέπει να στοχαστούμε και θα πρέπει να εφεύρουμε μέτρα που θα υποβοηθήσουν τους αλληλείς στο να έχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα στην άσκηση του επαγγελματός τους. Απασχόληση στον τομέα της αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Ο τομέας της αλληλείας, συμπεριλαμβανομένης και της υδατοκαλλιέργειας, εξακολουθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις να παράγει ετήσια εισοδήματα ύψους 34,2 δις ευρώ και δημιουργεί πάνω από 350.000 θέσεις εργασίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τομείς τη αλληλεία και τη ενατοκαλλιέργειας θεωρούνται σημαντικές πηγές εμέσων και αμέσων θέσεων απασχόληση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία ο αλλιευτικό κλάδος έχασε 30% των θέσεων εργασίας του. Έχοντας 23 εκατομμύρια, περίπου δηλαδή το 10% του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού άτομα να είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να ενισχύσουμε την αποσχόληση στον τομέα της αλληλείας και της συντοτοκαλλιέργειας και να διοχετεύσουμε ανέργους προς τους τομείς αυτούς. Ο αλληλευτικός τομέας μπορεί να παραμείνει βιώσιμος και ανταγωνιστικός μόνον εάν στελεχωθεί από επαρκή αριθμό εργαζομένων με την κατάλληλη κατάρτιση και τις απαραίτητες δεξιότητες. Καλείται η Επιτροπή να προωθήσει κατάλληλα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης καθώς και να εξεταστούν μέτρα προκειμένου να γίνει ελκυστικότερος ο κλάδος, ιδιαίτερα για τους νέους και να μελετηθούν μέθοδοι προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι επενδύσεις στον κλάδο. Το εύρος της έκθεσης είναι πολύ μεγάλο. Και καθότι το μέγεθος του κειμένου είναι περιορισμένο, προσπάθησα να επικεντρωθώ στα σημαντικά στοιχεία στα οποία αναφέρεται η ανακοίνωση της Επιτροπής. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για την πολύτιμη συμβολή τους μέσα από τη διατύπωση ιδεών και προτάσεων που διατυπώθηκαν είτε κατά την διάρκεια των συναντήσεων της Επιτροπής είτε σε ακροάσεις που διοργανώθηκαν. Οι τροπολογίες και προτάσεις από τους συναδέλφους μου είναι καλοδεχούμενες καθώς σκοπός είναι να παρουσιάσουμε μια κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα χαρώ να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαβράκο. Ο κύριος Κούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαβράκο για το γεγονός ότι πήρε και την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό σε σχέση με τη γενική κοινοποίηση για την μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε μια συνολική εικόνα για τη μεταρρύθμιση αυτή. Βέβαια είναι μια έκθεση πρωτοβουλία, αλλά μας δίνει την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων. Ο στόχος θα είναι να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με το πιο αποδοτικό τρόπο τους θαλάσσιους πόρους και φυσικά με τον πιο αηφόρο τρόπο και επομένως να διατηρήσουμε την ικανότητα αναπαραγωγής της βιομάζας στην ε, θάλασσα. Αυτό σημαίνει πρέπει να υπάρχει κάποια ασφάλεια στο σχεδιασμό μας, ότι θα πρέπει να έχουμε πολυετή σχέδια διαχείρισης για τα διάφορα αλλιευτικά είδη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία σε σχέση με τα αποθέματα αυτά, αλλά και συνεργασία με τα περιφερειακά αλλιευτικά συμβούλια, τα οποία μπορούν να προσφέρουν την ιδιαίτερη εμπειρία που έχουν στα θέματα αυτά. έχουμε και τις ε, μικρο, έχουμε <clears throat> μάλλον τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που λένε ότι υπάρχει υπεραλίευση και καταστρέφεται η βιολογική βάση της ε, αλίας. Αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε με την εμπειρία που έχουν και τη γνώση που έχουν τα περιφερειακά λιευτικά συμβούλια, τα ΡΑΚ. Δεν... Δεν πρέπει να παραμείνουμε λοιπόν μονάχα σε σενάρια αποκάλυψης για την αλληλευτική πολιτική το ένα σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει επίσης είναι πώς αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν τα ΑΤΑΚ, τα συνολικά αλλιεύματα, και πώς αυτά τα συνολικά αλλιεύματα δεν έχουν εξασφαλίσει την ε, βιωσιμότητα του τομέα. Πιστεύω όμως και πάλι και το επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς να έχουμε και τη γνώμη των αλλιών. Δεν μπορεί να αποφασίζεται η ποσόστοση για κάθε θαλάσσιο είδος με αυθαίρετο τρόπο από τον ένα χρόνο στον άλλο να αλλάζει άρδιν, χωρίς να ζητάμε τη γνώμη των αλλιέων. Επίσης για τους αλλιευτικούς στόλους. Η περιφερικοποίηση των μέτρων είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συλλογή στοιχείων για κάθε κράτος μέλος, για κάθε περιοχή πόσα σκάφη έχουν, πόσα μεγάλα είναι τα σκάφη, πόση ισχύ έχουν οι κινητήρες τους και κατά πόσο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αηφορία της αλίας σε κάθε περιφέρεια. Και επίσης και το, τα αλλιευτικά είδη, οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κάθε περιοχή, όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση που κάνουμε και είναι πολλοί από τους ε, βουλευτές μας που έρχονται από περιοχές μικρής και βιοτεχνικής αλίας και αυτοί μπορούν να μας δώσουν και τις δικές τους απόψεις. Επίσης για τα αλληλευτικά ε, έχουμε πολλές απώλειες από πτηνά όπως είναι η κορμοράνη, διάφορα αρπακτικά πτηνά τα οποία ε, οδηγούν σε απώλειες σε αυτά τα αλληλευτικά είδη. Σε άλλα αλλιευτικά είδη όμως έχει υπάρξει μια υπερ, ε, υπεράυξηση του πληθυσμού και δημιουργούν και πίεση στους ε, πόρους, στους διατροφικούς πόρους για τα άλλα θαλάσσια είδη. Και δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι και, αυτά θα πρέπει να υπόκειται σε μια διαδικασία προστασίας. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό σχέδιο διαχείρισης και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Η ηχθειοκαλλιέργεια επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα. Ξέρουμε από τις διάφορες έρευνες που έχουν λάβει χώρα τα προηγούμενα χρόνια ότι εμείς ως Ευρώπη με περίπου 8 εκατομμύρια τόνους αλλιευτικών προϊόντων είμαστε ο μεγαλύτερος καταναλωτής τέτοιων αλλιευτικών προϊόντων στον κόσμο, αλλά 70 με 80% από αυτά τα προϊόντα είναι εισαγωγές. Και επομένως εδώ είναι σημαντικό να σκεφτούμε και τα θέματα της προστασίας του καταναλωτή και την εφαρμογή των ίδιων κριτηρίων για τις εισαγωγές όπως αυτά τα οποία επιβάλλονται στους δικούς μας αλείς. Και πάλι επανέρχομαι στο θέμα της περιφερικοποίησης. Μέχρι ποιου βαθμού θα πρέπει να φτάσει η περιφερικοποίηση, μέχρι ποιου βαθμού θα πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες για ποσοστώσεις κτλ. Και φυσικά δεν πρέπει να αφήσουμε να επικεντρωθεί όλη αυτή η δραστηριότητα σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλους κεφαλαιοχικούς ομίλους. Θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα διατηρήσουμε και την επιβίωση των μικρών αλλιέων. Δεν θέλουμε οι μικροί αλλοίς τελικά να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, να πουλήσουν τα σκάφη τους και τις άδειέ τους και όλα αυτά να έρθουν στα χέρια μερικών μονάχα μεγάλων αλληλευτικών ομήλων. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σαλαβράκο γιατί ανέδειξε το θέμα αυτό και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε μέσα από τη συζήτηση να καταλήξουμε σε μια πιο συνεκτική πολιτική αλλιευτικών θεμάτων για το επόμενο διάστημα 2014-2020. Και σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αλίας και τις επενδύσεις, θέλουμε και εκεί να επιδοτήσουμε τη χρήση πιο αποδοτικών κινητήρων στα αλλιευτικά σκάφη, αλλά επίση να υποστηρίξουμε και την έρευνα στην ηχθειοκαλλιέργεια, να υπάρξουν επενδύσεις όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίσης και για δημόσια Ινστιτούτα τα οποία θα μπορούν να λειτουργήσουν στα κράτη-μέλη μας ως ερευνητικοί φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι την ε, θέση, τουλάχιστον από την άποψη οργάνωσης ε, του εγγράφου του συναδέλφου Σαλαβράκου. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία για αυτή την γνωμοδότηση συμπίπτει με μια σημαντική στιγμή διότι καλούμεθα να δώσουμε απαντήσεις σε, στα ερωτήματα αυτά σε σχέση με την μεταρρύθμιση εγώ θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω κάποιες σκέψεις. Θα ήθελα να... Εγώ θα έκανα κάποιες λιγότερες ερωτήσεις και κάποιες περισσότερες ε, ε, επιβεβαιώσεις ή διατυπώσεις. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να στραφούμε προς την Κομισιόν με μεγαλύτερη βεβαιότητα δηλαδή και όχι με τόσα πολλά ερωτήματα. Αν υπάρχει κάποιο όριο σήμερα στην κοινή αλληλευτική πολιτική, καθώς και στις προτάσεις ε, που συμπεριλαμβάνονται σε άλλες εκθέσεις. Αυτό το όριο είναι ότι πάντα μιλάμε για τα ίδια επιχειρήματα, προσπαθώντας να στοχεύσουμε καλύτερα για τα δίχτυα, για τον αριθμό των σκαφών, τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ακόμα στη συζήτηση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο κάτι το οποίο να μας υποδεικνύει τον δρόμο έτσι ώστε σε 5-10 χρόνια να μην είμαστε ακόμα εδώ και να μην συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα με κάποια λιγότερα αριθμητικά στοιχεία και μεγαλύτερες ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση των αποθεμάτων και την κατάσταση των αλλιών. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εμείς συμπληρωματικά ως Ευρώπη, δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας κάνουν να βλέπουμε μια θετική προοπτική. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα έγγραφο του Κοινοβουλίου θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τολμήσουμε να κάνουμε κάποιες περισσότερες υποδείξεις ή να δώσουμε προσανατολισμούς. Αν έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση έτσι όπως μας ε, προτείνεται, δεν ξέρω τελικά ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα στο τέλος της μεταρρύθμισης. Εγώ πιστεύω πως το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό. Δεν θα ήταν χρήσιμο ούτε για τον θάλασσα, ούτε για τα λιευτικά αποθέματα, ούτε και για τους αλείς. Κατά τη γνώμη μου πρέπει δηλαδή σε αυτό το έγγραφο να ενταχθούν κάποιες αρχές καθώς πρόκειται για ένα έγγραφο πρωτοβουλίας του ίδιου του Κοινοβουλίου και είναι χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα και να αλλάξει το σενάριο της οικονομίας αλλά και της ανάγκης ανασύστασης των αποθεμάτων. Εδώ και καιρό λέω ότι από αυτή τη μεταρρύθμιση λείπει η θάλασσα. Δεν υπάρχουν δράσεις για την θάλασσα ως, ως ένα μέσο ώστε να αντιστραφούν οι τάσεις. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με το περιεχόμενο, αλλά όχι με το δοχείο, που, τη θάλασσα που περιλαμβάνει όλες αυτές, όλα αυτά τα, τα θέματα. Πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο. Ποιες θα είναι οι πολιτικές για την ανασύσταση των αποθεμάτων, όχι ο περιορισμός των, της αλίευσης. Ποιες ε, δράσεις θα κάνουμε συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση που είναι η σταδιακή διαρθρωτική μείωση. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία, δεν οφείλεται στην αλία μόνο. Πρόκειται για μια διαρθρωτική μείωση των ε, αλλιευμάτων. Εάν δεν κάνουμε τέτοιου είδου προτάσει, δεν θα υπάρξει τίποτα που θα σταθεί. Δεν θα σταθούν ούτε τα δικαιώματα, ούτε τα μεγαλύτερα δίχτυα, ούτε η μείωση των σκαφών, ούτε η μείωση των ποσοστώσεων. Γιατί με κάθε μείωση των ποσοστώσεων θα γίνονται ε, περισσότεροι παράνομη αλληλεία. Πραγματικά λοιπόν πρέπει νομίζω να ανατρέψουμε την άποψή μας δεν ξέρω, αλλά θαραλέες επιλογές ε, κάποιο είδους, αλλά ξέρω και πέρα από αυτά που μπορεί να πω και που μπορεί να σας φανούν πολύ επαναστατικά εντός εισαγωγικών, αλλά να υποδείξουμε έναν στόχο όπου σημαντικές περιοχές της Ευρώπης θα γίνουν no fishing area, δηλαδή ε, περιοχές όπου δεν μπορεί κανείς να ψαρεύει, όχι για ένα-δυο μήνες μόνο, δηλαδή μόνο για την ε, βιολογική ανάπαυση, αλλά για κάποια χρόνια, μέχρι ότου η φύση να, το να επιτρέψει την ανασύσταση. Ή, εν περιπτώσει, να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις μέσω των οποίων εμείς να παίξουμε ένα ρόλο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ένα ρόλο τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε αναλάβει. Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να ορίζουμε κανόνες και εγώ σας αναφέρω την εμπειρία της Μεσογείου γιατί δεν παρενέβαινε προηγουμένω στην έκθεση της συναδέλφου Ρόσμπαχ γιατί Εκεί γινόταν λόγος για κάτι το διαφορετικό. Αλλά γιατί στη Μεσόγειο η κατάσταση είναι δραματική. Η εφαρμογή αυτού του κανονισμού είναι μηδενική. Μόνο αρνητικά στοιχεία έχουν, ε, έχει φέρει στην Αλία. Και το πολύ δραματικό είναι ότι τα δύο τρίτα του, της Μεσογείου δεν είναι καν ευρωπαϊκά. Εφόσον τα, στα δύο τρίτα της Μεσογείου αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται, ε, τότε δεν τίθεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν εγώ δεν αρκούμε σε αυτή τη φράση που λέει ότι η Κομισιόν που λέει, μπορεί να μας πει ποια μέτρα είναι αυτά που, που έχει αναλάβει ώστε να διασφαλίσει την υπεύθυνη και βιώσιμη αλληλεία. Εγώ θα ήθελα το Κοινοβούλιο να πει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλληλευτικών συμφωνιών στη Μεσόγειο που δεν θα σχετίζεται με το αλληλεύματα τα ΤΑΚ αλλά με, που θα σχετίζεται με τους ίδιους κανόνες γιατί είναι αυτή η κλειστή θάλασσα όπως είπαμε στην προηγούμενη παρέμβαση θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πούμε ότι πρέπει καταρχήν να αναζητήσουμε μια κοινή πολιτική και να τη στηρίξουμε. Τώρα ίσως θα γίνει αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες στη συζήτηση όταν θα μιλήσουμε για την εξωτερική μας πολιτική και για τις σχέσεις με τις χώρες τις υπόλοιπες. Αλλά αυτή η πρωτοβουλία μας μπορεί να εμπλουτιστεί κατά τη γνώμη μου προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω γιατί και έχω και άλλα να πω για την υδατοκαλλιέργεια κτλ. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτή η ιδέα να σας μεταφέρω. Ότι δηλαδή πρέπει να βάλουμε εδώ την θάλασσα ως το μέρος όπου θα πρέπει να οικοδομήσουμε πολιτικές και να βρούμε ένα σύστημα μέσω των διεθνών μας σχέσεων να μην ασχολούμαστε μόνο με τις ε, συμβάσεις ε, σε διεθνές επίπεδο, σε διεθνή βήματα, γιατί αυτές χρυσό του να οριστούν και να εφαρμοστούν θα έχουμε νεκρή θάλασσα. Θα έχει επεκταθεί η νεκρή θάλασσα και στην Μεσόγειο και στην ε, Μαύρη θάλασσα. Η νεκρή θάλασσα είναι εκείνη εκεί μετά από την Ιορδανία. Αλλά θα έχει γίνει νεκρή και η Μαύρη Θάλασσα και η Μεσόγειος μέχρι ότου να εφαρμόσουν όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν και θα ασχοληθώ με αυτό μέχρι που να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις τροπολογίες και θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για αυτά τα θέματα. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω και τη γνώμη των συναδέλφων για αυτό το θέμα, γιατί κατά τη γνώμη μου με κάποια ελαφρότητα μιλάμε για μια πολιτική που βασίζεται στις ίδιες προϋποθέσεις, στους ίδιους όρους. Θα πρέπει να σκεφτούμε νέες υποθέσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Λόβεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σαλαβράκο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή έκθεση και περιλαμβάνονται διάφορα καλά σημεία με τα οποία συμφωνούμε Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Να αναφερθούμε στο ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα αποθέματα σε ένα επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε αυτό το above στα αγγλικά πάνω, δηλαδή από το επίπεδο αυτό του MSY. Ο κύριος Αλαβράκος πολλές φορές λέει στην εκθεσή του ότι χρειαζόμαστε επιστημονικά δεδομένα, επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν όμως έχουμε αποθέματα σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε εξασφαλισμένοι δηλαδή σε ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τότε κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Είμαστε πιο εξασφαλισμένοι ουσιαστικά. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε κάθε ψάρι στη θάλασσα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα αποθέματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα, μια ζώνη ευελιξία, ασφάλεια, προκειμένου να είμαστε εξασφαλισμένοι. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αλληλευτικά αποθέματα υψηλότερα από το επίπεδο που απαιτείται για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν θέλουμε, όπως είπε ο κύριος Μιλάν, να αναλάβουμε υπόψη μας τα οικοσυστήματα και το πώς ε, ουσιαστικά λειτουργεί η θάλασσα και οι ωκεανοί, αν, έχουμε απλώς, αν περιοριστούμε απλώς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ουσιαστικά κινούμαστε με μια λογική αλίευσης, αλίας. Προσεγγίσουμε μόνο κατά αυτόν τον τρόπο τη θάλασσα και τους ωκεανούς βλέποντας ουσιαστικά ποια ποσότητα μπορούμε να βγάλουμε, να ψαρέψουμε μέσα στη θάλασσα. Αν θέλουμε όμως να έχουμε μια οικοσυστημική προσέγγιση, τότε θα πρέπει να έχουμε υψηλότερα αποθέματα, να προβλέψουμε ένα υψηλότερο επίπεδο για τα αποθέματα. Ο κ. Σαλαβράκος επίσης πολλές φορές αναφέρθηκε στο ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια οικονομική βοήθεια προς τις κοινότητες εκείνες οι οποίες ε, επηρεάζονται και θα επηρεαστούν από περισσότερες περικοπές στην απασχόληση και το καθεξής. Συμφωνώ είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης. Θα πρέπει να δοθεί μια προστιθέμενη αξία σε συγκεκριμένου τομείς των στόλων. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας στην έκθεση αυτή από το New Economic Foundation. Η έκθεση εδώ πέρα έχει τον τίτλο θέσεις απασχόλησης που χάνονται στη θάλασσα. Οι επιστήμονες λοιπόν του Ιδρύματος αυτού κάνανε μια πολύ απλή άσκηση. Αυτό που κάνανε είναι ότι υπολογίσανε τους, τα, 20, τα 43 σημαντικότερα εμπορικά αποθέματα παγκοσμίω. Θέλησαν ουσιαστικά να, δούσουν, να, να δούνε ποια είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορούμε να έχουμε για τα αποθέματα αυτά. και είδανε ότι υπήρχε δυνατότητα για ένα επιπλέον 33% σε σχέση με τα προβλεπόμενα επίπεδα. Και η επιπρόσθετη αξία είναι 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Και οι θέσει απασχόλησης που μπορούν να δημιουργηθούν είναι 100.000 θέσεις απασχόλησης. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για μέγιστη βιώσιμη απόδοση, έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει ε, να κάνουμε περικοπές, ότι πρέπει να κάνουμε μειώσεις. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι ε, αν θέλουμε ως πολιτικοί να προστατεύσουμε και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, και ξέρετε ότι διανύουμε μια οικονομική κρίση που θέλουμε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια τη οποία θέλουμε να περασπιστούμε και τι θέσει απασχόληση. Αν θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό στην Αλία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν καταφέρουμε να έχουμε αποθέματα που θα είναι αρκετά πιο ψηλά από, αυτά που απαιτούνται για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Επίση, ε, διαφορετικά ληφτικά μέσα, εργαλεία επηρεάζουν και με διαφορετικό τρόπο τις θέσεις απασχόλησης. Αν βέβαια χρησιμοποιήσουμε τα υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητα, αυτό θα οδηγήσει και σε χαμηλότερε θέσει εργασία και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο κύριο Σαλαμπράκο αναφέρθηκε επίση στα καύσιμα και στην αυξανόμενη τιμή των καυσίμων. Όλε οι μελέτε που έχουν γίνει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν ότι το τμήμα του στόλου που πειράζεται περισσότερο από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων είναι οι στόλοι οι οποίοι είναι λιγότερο φιλικοί προς το περιβάλλον. Επομένως, οι στόλοι της μικρής ε, αλίας, της αλίας μικρής κλίμακος, επηρεάζονται λιγότερο από αυτές τις απότομες αυξήσεις στα καύσιμα. Με το να έχουμε επίσης αποθέματα πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, έχουμε λιγότερη ανάγκη για να χρησιμοποιήσουμε καύσιμα. Ουσιαστικά ο Αλιεύς ε, με το σκάφος του δεν χρειάζεται να περάσει τόση πολλή ώρα στα νυχτά της θάλασσας. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε το γρηγορότερο δυνατό να ανακτήσουμε τα αποθέματα πάνω από το MSY, πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο, δίνοντας επίσης λιγότερες επιδοτήσεις και λιγότερη οικονομική υποστήριξη. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Μιλάνα όσον αφορά, τις, ε, όσον αφορά την προστασία των θαλασσών είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια της πολιτικής αλίας να ασχοληθούμε και με την ίδια την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και παντού στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα τα δεδομένα, Ο κ. Σαλαβράκο μα είπε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να διαβιβάζουν περισσότερα δεδομένα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν αν δεν δίνουν τα απαραίτητα δεδομένα. Και αυτό γίνεται τώρα. Δεν διαβιβάζουν τα απαραίτητα δεδομένα και αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να προβλέπονται λοιπόν κυρώσει. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ε, χρηματοοικονομική υποστήριξη και δεν θα πρέπει να έχουν καν πρόσβαση στου ελευτικού πόρου εν τέλει, αν δεν δίνουν αυτά τα απαραίτητα δεδομένα κύριος Ντέβις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο και εγώ θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και να τονίσω ότι έκανε μια ρεαλιστική και ισορροπημένη και προοδευτική έκθεση ο εισηγητής, κάτι το οποίο με χαροποιεί. Για να σας δώσω ένα δείγμα αυτής της ε, ισορροπίας, αναφέρει ο, ο κύριος Σίτης. τις ε, ανησυχίες του για τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Εγώ εργάστηκα για τις τροπολογίες σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση τη Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα θέματα αυτά. Όλα τα κόμματα, με τη δική μου εξαίρεση ίσως, θέλανε να μετακινηθούν από την υποχρεωτική εφαρμογή των μεταβιβάσιων ποσοστώσεων σε προαιρετική ε, χρήση μεταφερόμενων ποσοστώσεων. Αλλιώ πρέπει να μειώσουμε την αλληλευτική ικανότητα. Αλλά πώ θα το κάνουμε αυτό. Γιατί τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να είχαν μειώσει την αλληλευτική ικανότητα εάν το θέλαν. Δεν το θέλουν. Όμω και αυτό έχουν δείξει. Για την περιφερειοποίηση είναι λογικό αυτό που λέει ο εισηγητή. Λέει ότι δεν υπάρχουν. Ξέρουμε όλοι ότι ο Γενικό Κανονισμό δεν λέει πολλά πράγματα για την περιφερειοποίηση. Ο κ. Σαλαβράκη τονίζει ότι πρέπει να είναι εκ των κάτω προ τα άνω. Έτσι τα περιφερειακά συμβουλία τα ΡΑΚ θα πρέπει να λειτουργήσουν και να πάρουν την πρωτοβουλία στα θέματα αυτά με προτάσεις. Για τις απορρίψεις. Ναι, καταρχήν είναι κάτι το απαράδεκτο. Ισμαήλ λένε ότι είναι και ανήθικο αυτό. 1,7 εκατομμύρια τόνοι ε, βρόσιμων ψαριών τα οποία απορρίπτονται κάθε χρόνο. Οι Σκοτσέζοι συνάδελφοι μπορούν να το αναφέρουν αυτό ίσως και να επιβεβαιώσουμε, υπήρξε ένα, ένα πείραμα με το να εκφορτώνονται όλα τα ψάρια και χρήση επιλεκτικών ειδών αλίας και αυτό μείωσε σημαντικά τις παράλληλες αλίες. Έχει ξεπεράσει καν και τις προσδοκίες των αλιέων αυτό το νέο πείραμα. Παρά το ότι δεν μπορεί να γίνει παντού κάτι τέτοιο, δείχνει αυτό ότι το να είναι υποχρεωτικό όλα τα ήδη τα θαλάσσια που αλλιεύονται να εκφορτώνονται, αυτό δίνει κίνητρα για να έχει κανείς πιο επιλεκτική αλληλεία, κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί αρκετά γρήγορο και έτσι δίνει κίνητρα στους αλλιεί να μειώσουν, να την, τα παράλληλα αλλιεύματα, τα παρά, παράπλευρα αλλιεύματα. Το θέμα των μικρών αλλιέων επίσης είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι να το υποστηρίξουμε, αλλά αυτό είναι μια ευθύνη των κρατών μελών σε κύριο επίπεδο. Γιατί οι αλληλευτικές ευκαιρίες δίνονται στα κράτη-μέλη και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για την κατανομή του. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη και ένα από αυτά είναι το δικό μου που δεν βοηθούν ιδιαίτερα του μικρού αλείς. Περίπου 4% των συνολικών αλληλευτικών ευκαιριών που δεν είναι ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουμε την ευμάρεια των μικρών αλλιών. Τέλος, να πω κάτι για τα σχόλια του κυρίου Μιλάν. Γιατί ήταν κάπως αποκαλυπτικά αυτά που είπε σε ό,τι αφορά την κατάρρευση των αλληλευτικών πόρων. Πιο πολύ και από αυτά τα οποία λέω εγώ, πιο μεγάλο κίνδυνο διέγραψε από αυτά που λέω εγώ. Και σωστό είναι να έχουμε περισσότερα ψάρια και να υπάρξει διατήρησή τους. Αλλά είπατε κύριε Μιλάνα ότι θεωρείτε ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική και ο αντίστοιχο κανονισμός δεν θα βοηθήσουν την ανάκαμψη των βιολογικών πόρων. Ήσασταν τελείως αρνητικός. Φοβηθήκατε ότι μια μείωση των ποσοστώσεων θα οδηγούσε σε πιο πολύ παράνομη και εκτός ελέγχου αλία. Εγώ πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσουμε πολιτική βούληση μπορούμε να μειώσουμε την παράτυπη και παράνομη αλία. Στη Σκωτία ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκφορτώναν παράνομα ψάρια αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Πάλι οι Σκότοι, οι συνάδελφοί μου, μπορούν εδώ να με διαψεύσουν αν θέλουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέω ευσταθεί. Μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο κανονισμός που εγκρίναμε τον Ιούλιο λέει ότι πρέπει να, ξαναφύγουμε, πια από μια κοντόφθαλμη οπτική, να αποφασίζουν κάθε Δεκέμβριο οι Υπουργοί Αλίας ποιες είναι οι ποσοστώσεις, και να κινηθούμε προς ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο προγραμματικής και όταν τα κρατημέλη δεν κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν κυρώσει. και να μπορέσουμε να έχουμε σωστούς στόχους και φυσικά να σταματήσουμε και τις απορρίψεις. Και εγώ μπορώ να είμαι απεσιόδοξο. <clears throat> Δεν πιστεύω ότι αν αυτά τα κύρια στοιχεία, τα κέρια στοιχεία είναι στον κανονισμό, αυτό θα μπορούσε να χειροτερέψει περισσότερο την κατάσταση. Νομίζω ότι απλώς θα τη βελτιώσει. Ευχαριστώ κύριε Ντέβιτ. Ο κύριος Χότον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο εισηγητής συνέταξε μια πολύ σφαιρική, πλήρη έκθεση. Θα επικεντρωθώ στα σημεία αυτά με τα οποία συμφωνώ. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε και να τα υποστηρίξουμε επίση και στον, στην έκθεση που έχουμε για τον βασικό κανονισμό. Η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική σε διάφορες από τις παραγράφους της έκθεσης. Θα ακολουθήσω τη σειρά που έχει και έκθεση. Μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ιδίως όταν έχουμε μεικτή αλία. Είναι καλό να έχουμε στόχους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι και ρεαλιστικοί και θα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας. Βέβαια, ορισμένες φορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποιες ιδιαίτερες ε, ε, πραγματικότητες, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οι απορρίψεις. Ξέρετε ότι οι απορρίψεις είναι ένα σκάνδαλο πραγματικά όταν έχουμε αλλιεύματα τα οποία απλώς εκφορτώνονται στη θάλασσα, απορρίπτονται στη θάλασσα Και όντως εδώ πέρα θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αποφύγουμε καταρχάς τα ανεπιθύμητα αλλιεύματα, τα ανεπιθύμητα παρεπίπτοντα αλλιεύματα, προκειμένου να μην καταλήγουμε στο φαινόμενο αυτό της απόρριψης. Έχουν γίνει όμως πολλές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε και το όλο πρόγραμμα εκφόρτωσης και αποθήκευσης των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. Ξέρετε ότι θα πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες χρόνος και θα πρέπει να έχουμε και ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα προκειμένου να εξαλείψουμε τελικά τις απορρίψεις και όχι απλώς μία απαγόρευση. Αργότερα στην εκθεσή του, ο κύριος εισηγητής λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα. Και ο κύριος Ντέιβις πολύ σωστά μας είπε ότι υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα εν εξελίξη που δείχνουν τελικά όντως οδηγούμαστε σε μείωση των απορρίψεων. Δεν είναι μόνο η απειλή της απαγόρευσης που έχει φέρει το αποτέλεσμα αυτό, είναι ότι έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα. όπως για παράδειγμα επιπλέον δυνατότητα λιευτικής προσπάθειας στη θάλασσα, επιπλέον μέρες για ορισμένα σκάφη, για παράδειγμα στη Σκοτία, τα οποία σε θελούσια βάση συνεργάζονται στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα επιτυχώς. Θα ήθελα λοιπόν όχι απλώς να ενθαρρύνουμε νέα πιλωτικά προγράμματα, αλλά να δούμε και τι γίνεται ήδη και πώς τελικά θα καταφέρουμε να επιβραπεύσουμε και όχι να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές αυτές. Και δεν θα πρέπει να είναι το μόνο μέσο το οποίο προτείνεται για την μείωση της πλεονάζουσας αλλιευτικής ικανότητας. Πρέπει να δούμε ότι σε ορισμένες αλλιευτικές χώρες, περιοχές όπως η δικιά μου η Σκωτία, ήδη είχαμε υποχρεωτική καταστροφή ορισμένων σκαφών και βέβαια αυτό οδήγησε σε μείωση θέσεων απασχόλησης την τελευταία αυτή δεκαετία. Και σε αντάλλαγμα τώρα πρέπει να μας πούν ότι θα έχουμε μεταβιβάσιμε ελευτικέ παραχωρήσεις. Και όπως λέμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εγγραφό τη, αυτέ οι παραχωρήσεις μπορούν να πάρουν και διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό όμως θα οδηγήσει μόνο σε συγκέντρωση τελικά της δραστηριότητας και αυτό θα ήταν καταστροφικό για πολλές παράκτιες κοινότητες. Και γι' αυτό το λόγο τελικά οι μεταβιβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της αλληλευτικής ικανότητας. Γιατί ουσιαστικά οι πολύ απότομες αλλαγές στην αγορά οδηγούν τελικά σε συγκέντρωση της δραστηριότητας, αλληλευτικής δραστηριότητας. Και βέβαια έχουμε και μια συγκέντρωση της όλης δραστηριότητας στην γη, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες εκφόρτωσης κτλ. Δεν νομίζω πάντως ότι έχουν προβλεφθεί ακόμα τα απαραίτητα ειχέγγια για το σύστημα αυτό και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο εισηγητή πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τον κοινωνικο-οικονομικό τομέα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτική πολιτικής. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διατήρηση και η βιωσιμότητα των κοινοτήτων που ζουν από την αλία καθώς επίσης και η συντήρηση προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Και ξέρετε ότι όλα τα δύο αυτά στοιχεία αλληλοεξαρτώνται τελικά. Αυτοί που έχουν να κερδίσουν περισσότερο από τις πολιτικές συντήρησης του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι ουσιαστικά οι αλλιευτικές κοινότητες οι οποίες εξαρτώνται από το θαλάσσιο αυτό περιβάλλον. Και η κοινή αλλιευτική πολιτική μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Κάποιοι λύθοι κανόνες πολλές φορές προτείνονται και ουσιαστικά περιοριζόμαστε μόνο σε κάποιους φόρους και σε κάποιες ποσοστώσεις. Και το μόνο που έχουμε καταφέρει τελικά είναι να έχουμε πολύ χαμηλές ποσοστώσεις που ουσιαστικά αποτελούν λόγο για τον οποίο έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο εκφορτώσεων. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική αυτή. Και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, περιφερειοποίηση. Εγώ θα ήθελα να έχουμε και τον όρο αποκέντρωση. Είναι σημαντικό να έχουμε την αποκέντρωση και ως πρώτη προτεραιότητά μας στην έκθεση αυτή. Τα όσα είπα σήμερα θα καταφέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα αν κάποιες αποφάσεις διαχείρισης μπορούν να ληφθούν σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο και αν μπορούν να έχουν σημαντικότερο λόγο οι ίδιες ηλεκτρικές κοινότητες, οι χώρες αυτές οι οποίες εξαρτώνται πολύ περισσότερο από την αλία. Αυτές θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά για το αν θα επιβιώσουν ή για το αν θα, αποφύγουν, αν θα αποτύχουν τελικά στο να επιβιώσουν. Νομίζω ότι το σημαντικότερο κίνητρο που μπορούμε να δώσουμε είναι την δυνατότητα να εγκρίνονται τέτοια μέτρα διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα επηρεάσει θετικά την κοινή ελευτική πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Φερέιρα. Χωρίς μικρόφωνο. Αμικρόφωνος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Ορισμένα σύντομα σχόλια μονάχα για ορισμένα από τα ζητήματα που ηγέθησαν εδώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι πρόκειται για μια έκθεση που αφορά τη γενική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μια τέτοια έκθεση που αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή για την οποία είναι γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, ακόμα και διαμετρικά αντίθετες, αυτό απαιτεί από τον εισηγητή και κάποια πολιτική ευελιξία για να μπορέσει να εξασφαλίσει μια συνένεση και μια κατά κάποιο τρόπο συμφιλίωση αντίθετων απόψεων. Με όλη την προσοχή και την ε, ευελιξία και την ικανότητα που μπορεί να έχει ένας εισηγητής, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μονάχα εναλλακτικά σενάρια μπορεί κανείς να λάβει υπόψη. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλους, δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το θέμα των μεταφερομένων αλληλευτικών ποσοστώσεων. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση συνενετική. Δεν υπάρχει περιθώριο. Είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνει κανείς. Ορισμένοι θα ικανοποιηθούν, ορισμένοι όχι. Αυτό είναι το πρώτο σημείο λοιπόν που ήθελα να θίξω. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή στη γενική της μορφή μου φαίνεται ότι είναι πολύ ισορροπημένη. Περισσότερο ισορροπημένη από ότι και η ανακοίνωση της Κομισιόν. γιατί καλύπτει και τις τρεις διαστάσεις που θα πρέπει να έχει μια πολιτική αλίας. Την πολιτική του περιβάλλοντος, προφανώς, που είναι το πρώτο σημείο που εξηγείται, την οικονομική και την κοινωνική πτυχή που καλύπτονται και αυτές σε, σε οικία κεφάλαια. Αυτά είναι στοιχεία που η Κομισιόν δεν τα είχε λάβει ιδιαίτερα υπόψη ενώ στον, στην πρόταση του εισηγητή έχουν μεγαλύτερη ισορροπία, πιο ισορροπημένη θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το εξάρω και να το αναφέρω. Η Κομισιόν ξεκινά από την αρχή ότι εάν θέσει κάποιους στόχους περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όλοι οι άλλοι στόχοι που έχουν οικονομικό ή κοινωνικό χαρακτήρα με αυτόματο τρόπο θα επιτευχθούν, αλλά αυτό δεν είναι σωστό μπορούμε να έχουμε στόχους που θα αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι στόχοι μέσα σε μια πολιτική αλίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε τους οικονομικούς ή τους κοινωνικούς στόχους. Και επομένω νομίζω ότι υπήρχε αυτή η, αυτό το έλλειμμα στην πρόταση της που έχει καλυφθεί από τον εισηγητή. Για το πρώτο κεφάλαιο, για την βιωσιμότητα σε επίπεδο περιβάλλοντος, αναφέρθηκαν τα ζητήματα αυτά από τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που αναφέρει κάποια από αυτά ο εισηγητής, η βελτίωση της ε, επιλεκτικότητος στις μεθόδους αλίας, η ανάπτυξη νέων τεχνικών κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Όλα αυτά θα δώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Και αν μπορέσουμε να μειώσουμε τις απορρίψεις, κάτι το οποίο είναι σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει να λάβουμε και κάποια πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη <clears throat> την τεράστια απόσταση που υπάρχει μεταξύ της αλίας στον βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα λοιπόν από αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα έχω προτείνει και εγώ στην ε, έκθεση για τον κανονισμό της κοινή οργάνωσης αγοράς έχω αναφέρει και ορισμένα μέτρα τα οποία κατά την άποψή μου θα εγγυηθούν και θα υποστηρίξουν σε, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο την μείωση και την εξάλληψη των απορρίψεων. Δηλαδή να υπάρχει και μια ελάχιστη επιδότηση για το κόστος εκφόρτωσης των αλλιευμάτων. Η ιδέα των πιλωτικών σχεδίων μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Να αναπτύξουμε λοιπόν τέτοια σχέδια στο τομέα αυτό. Για την συλλογή δεδομένων τώρα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το βασικό είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις στις χώρες οι οποίες δεν συλλέγουν και δεν παρουσιάζουν δεδομένα. Λες και την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν ως εκθαύματος αυτά τα δεδομένα. Αλλά εγώ επιμένω, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πραγματικότητα που έχουμε στις χώρες μας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που έχουν πολύ διαφορετικές αρχικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τη συλλογή των δεδομένων. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει σαφής έλλειψη υποδομών και μέσων για να υπάρξει αυτή η συλλογή στοιχείων. Το υπογραμμίζω αυτό. Και εδώ υπάρχει και μια έλλειψη υπευθυνοποίηση τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινοτικού προπολογισμού. Κάνουμε τώρα μια σημαντική αλλαγή που έλαβε χώρα με τη συνδίκη τη Λισαβόνα που οδήγησε στο ότι η διαχείριση των αλληλευτικών πόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι λαθασμένο κατά την άποψή μου, αλλά αυτό λέει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά η μέγιστη χρηματοδότηση που δίνει η Κομισιόν στα κράτη-μέλη για να συλλέγονται στοιχεία είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 50% όπως και πριν από τη θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει περισσότερο λοιπόν από τα θέματα από το επίπεδο αυτό η Κομισιόν. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το ανώτατο επίπεδο και ίσως θα ήταν χρήσιμο και ο εισηγητής να θέσει αυτό το θέμα, διότι αναφέρεται στα ζητήματα των μέσων που είναι απαραίτητα, στην τεχνική αρρωγή και την οικονομική αρρωγή της Κομισιόν και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να αυξήσουμε τη μέγιστη συγχρηματοδότηση που αυτή τη στιγμή είναι 50% για την συλλογή στοιχείων. Τώρα, τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα των μεταφερομένων ποσοστώσεων. Εδώ πιστεύω πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ προτάσεις. Και οι προτάσεις που έχουμε, είτε ένα, σύντομο, ένα, συγγνώμη, σύστημα το οποίο είναι υποχρεωτικό, όπως ζητάει η Κομισιόν, ή ένα εθελοντικό. Δεν υπάρχει μέσο έδαφος. Εδώ μπορούμε να σκεφτούμε όμως ένα σύστημα που θα είναι υποχρεωτικό αυτό το καθεστώς, εκτός αν το κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέτρα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο. Εγώ ανέφερα προηγουμένως λόγους για τους οποίους δεν θέλω να είναι υποχρεωτικό το σύστημα αυτό. Μπορούμε να επανέλθουμε στην επόμενη, στις επόμενες εκθέσεις. Θα πρέπει όμως να πούμε, εάν θέλουμε να είναι εθελοντικό, ότι θα είναι εθελοντικό και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό το να προσπαθήσουμε να συμβιβάσουμε τις δύο αυτές αντίθετες απόψεις δεν μου φαίνεται ότι ευσταθεί γιατί πολλές από τις ε, υποθέσεις που βρίσκονται πίσω από το σενάριο των μεταφορμένων ποσοστώσεων δεν έχουν κάποια επιστημονική βάση. Θα πρέπει να έχουμε κάποια εμπειρικά στοιχεία που να μας δείξουν ότι αυτό το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να έχουμε καλύτερες διασφαλίσεις από αυτές που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Δεν πρέπει λοιπόν να ε, επιμείνω γι' αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν και ρήτρες διασφάλισης. Και γι' αυτό υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σύστημα αυτό. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο εδώ να είναι πιο σαφής η έκθεση του εισηγητή. Επίσης, για μένα είναι θετικά όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της απασχόλησης, η υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η καλύτερη κατάρτιση των αλλιέων, η ιδιαιτερότητα της μικρής και βιοτεχνικής αλλαγίας που αναφέρει ο Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία τα βρίσκω πολύ Περιφερικοποίηση. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. Θα ήθελα να είναι, είναι πιο εκτενής η έκθεση για τα θέματα περιφερικοποίησης γιατί και εδώ είναι ένας τομέας όπου η πρόταση της Κομισιόν ε, μακρηγορεί. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε έμφαση στη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα θέματα για, τα, για τις αποκλειστικές περιοχές αλίας των 12 αλιών, όλ, ε, όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν σε περιφερειακό επίπεδο και θα ήθελα και μέσα στην Επιτροπή μας να μπορέσουμε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Φεραίρα. Κύριος Παντεκούπερ από την Κομισιόν. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας και συγχαρώντας τον ε, εισηγητή για την έκθεση αυτή. Είναι ιδιαίτερα πλήρης η έκθεση αλλά και σύντομη παράλληλα. Δηλαδή αναφέρεται στα περισσότερα σημεία το οποία αναφέρουμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας. Με τρόπο ιδιαίτερα ευσύνοπτο. Πέρα από αυτά, είμαστε υπέρ της ε, έκθεσης, επί της αρχής είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη, δεν συμφωνούμε απαραίτητα με κάθε παράγραφο ή κάθε λέξη που χρησιμοποιείται στην έκθεση, ωστόσο θεωρούμε ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση, μια ισορροπημένη απάντηση μάλλον στην ανακοίνωσή μας. Να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Πολύ σωστά, ο εισηγητής λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα, δύο από τα σημαντικότερα σημεία στην πολιτική διατήρησης, συντήρησης, είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση και ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτήν το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μία προθεσμία, επομένως υπάρχει μία υποστήριξη της έκθεσης για την προσέγγιση αυτή της Επιτροπής. Επίσης, συμφωνούμε με τα όσα λέγονται για τις απορρίψεις. Όντως θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ στα πλαίσια της πολιτικής ε, για την εξάλληψη των απορρίψεων. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί και με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό πρόγραμμα. Πρέπει επίσης να δούμε και ποιες υποχρεώσεις θα υπάρχουν για την εκφόρτωση. Ασχολούμαστε πάντως με όλες αυτές τις προτάσεις που γίνονται στην έκθεσή σας. Ξέρουμε όμως ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον ελευτικό κλάδο. Και συμφωνούμε πάντως με τα όσα λέγονται για τις απορρίψεις και θεωρούμε ότι μέσω των παραγράφων αυτών υποστηρίζει ουσιαστικά και την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνουμε επίσης τα σχόλια τα οποία έγιναν και στην έκθεση αλλά και στη συζήτηση όσον αφορά την κοινοοικονομική βιωσιμότητα και εμείς αυτό προσπαθούμε να πούμε στην έκθεσή μας. Η ε, κοινωνικονομική βιωσιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς αντιμετωπίζουμε τους στόλους, αλλά και τι κάνουμε για τις ε, παράκτιες κοινότητες όχι τόσο στο βασικό κανονισμό, όσο στην ε, πρόταση για το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εκφράσουμε εκεί, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τις ε, αλλιευτικές παράκτιες κοινότητες. Επίσης εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που έχει καταβάλει ο εισηγητής όταν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της συλλογής των δεδομένων καθώς επίσης και στην απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη που πρέπει να υπάρχει για τον ελευτικό τομέα. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό για την πολιτική μας και ό,τι προσπαθούμε να σημειώνουμε συνεχώς πρόοδο, υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση σημαντικό και πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων όχι μόνο από τα κράτη-μέλη αλλά και από τους ίδιους τους αλείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει λοιπόν κάθε σχετική προσπάθεια. Θεωρούμε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό και απαντά εδώ σε μία από τις παρεμβάσεις που γίνανε. Επί του παρόντο, τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν καν τα απαραίτητα διαθέσιμα ποσά που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο για την συλλογή των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τι προσπάθειε και στη διαβούλευση και στην εταιρική σχέση που έχουμε με τον αλληλευτικό κλάδο, γιατί πολλά από τα στοιχεία έρχονται τελικά από τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο. Ευχαριστούμε πάντως την εισηγητή που ανεφέρθηκε στο σημείο αυτό. Όσον αφορά τώρα την περιφερειοποίηση. Μόλις έχουμε δεχθεί επικρίσεις, θεωρούμε ότι κάνουμε μια πολύ δυναμική πρόταση όσον αφορά την περιφερειοποίηση. Ξέρετε ότι η συνθήκη επιτρέπει συγκεκριμένες μόνο μεθόδους. Εμείς όμως έχουμε κάνει μια πολύ δυναμική παρουσίαση, πρόταση με συγχωρείτε όσον αφορά την περιφερειοποίηση. Υπάρχει μια γενικότερη αναγνώριση για την ανάγκη της περιφερειοποίησης. Μπορούμε όμως να προσαρμόσουμε προφανώς την πρότασή μας αυτή σε οποιαδήποτε βελτιωμένη πρόταση μπορεί να έρθει από εσά. Πάντως στην ε, έκθεση του εισηγητή αναφέρονται όλα τα ζητήματα που άπτονται της περιφερειοποίησης, όπως τα περιφερειακά συμβούλια, η προσέγγιση ε, από τη βάση προς τα άνω και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, και το λέω ότι αποδεχόμαστε όλες τις προτάσεις που κάνει ο εισηγητή για την περιφερειοποίηση. Σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να εκφραστώ, να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή και την ομάδα του για την εξαιρετική αυτή δουλειά και προσβλέπουμε στι μελλοντικέ συζητήσει που θα γίνουν για την έκθεση αυτή. Κύριο Σαλαβράκο, για να κλείσει τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλου του συναδέλφου και τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν για τι θέσει του πάνω στην προσπάθεια που έκανα εγώ και η ομάδα μου και οι συνεργάτες μου. Ε, συμφωνώ με όλε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ωστόσο θα ήθελα να παρατηρήσω ότι από την εμπειρία μου σαν νομικού πιστεύω ότι η επιτυχία ενός νομοθετήματος βασίζεται στην εκτεταμένη αποδοχή και εφαρμογή του. Και πρέπει ένα νομοθέτημα να είναι δυναμικό και όχι στατικό. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει η σοβαρότητα του ελέγχου της εφαρμογής. Όλα αυτά τα πράγματα τα συνεκτίμησα διότι η γενική φιλοσοφία της εκθέσεως είναι μια πρόταση πλαίσιο που από την εμπειρία την οποία έχουμε σε σχέση με το πώς λειτουργούν τα κράτη παραδείγματο χάρη στο θέμα της ε, παραχωρήσεως στοιχείων μας δημιουργούνται επιφυλάξεις για την δυνατότητα της πλήρους εφαρμογής αν μπούμε σε πιο λεπτομεριακά μέτρα. Ε, λαμβάνω επίσης υπόψη ότι Βρισκόμαστε σε μια εποχή ε, που οικονομικά και κοινωνικά η Ευρώπη μετεξελίσσεται και θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και πρέπει να μην φυγούν αλλά απευθεία να δοθεί ιδιαίτερα έμφαση στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους και τους επικείμενους Ευρωπαίους. Διότι, εάν δούμε τα στοιχεία, η Ευρώπη του σήμερα είναι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού και παράγει το 32% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Ευρώπη του 2030 θα είναι το 4-5% του παγκόσμιου πληθυσμού και θα παράγει δυστυχώς το 10 με 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Θέλουμε δεν θέλουμε, η Ευρώπη του 2030 θα έχει κατά 50% λιγότερους Ευρωπαίους. Εν τω μεταξύ θα έχουν γεννηθεί 600 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι προερχόμενοι από περιοχές μουσουλμανικής επιρροής. Και δεν έχω τίποτα βέβαια με τις θρησκείες. Απλώς το λέω για να δούμε τι γίνεται γύρω μας και πώς νομοθετούμε και πού θα διοχετεύσουμε όλο αυτό το πλήθος. Άρα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να συντηρήσουμε τις θέσεις εργασίας όσες υπάρχουν στην Ευρώπη και να τις επαυξήσουμε. Και ιδιαίτερα σε επίπεδο που δεν χρειάζονται σπουδαιότατες ειδικέ γνώσεις όπως είναι η αλληλεία και μπορεί να γίνει ευρεία προσαρμογή και μη μορφωμένων πληθυσμών ούτως ώστε να αποκτήσουν τις ιδιότητες για να είναι, γίνουν καλοί αλληλείς. Στις αρχές της δικηγορίας μου τα πληρώματα των του ελληνικού στόλου που εξακολουθεί να είναι πρώτο στην ανθρωπότητα είναι ότι ήταν Έλληνες Σήμερα είναι Σομαλί. Δεν έχουμε κανένα Έλληνα εκεί. Δηλαδή όλα αυτά τα λαμβάνω υπόψη μου και παρακαλώ να τα λάβουν υπόψη τους και όλοι οι συνάδελφοι και δέχομαι όλους τους, όλους τους προβληματισμούς τους. Θέλω κι εγώ να είμαι δυναμικότερος και να βγάλουμε κάτι το πιο δυναμικό από αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει να είναι και εφαρμόσιμο και εφικτό. Εν πάση περιπτώσει, όσες ιδέες ακούστηκαν ήταν εξαιρετικές και καμία από αυτές δεν με βρίσκει ε, αντίθετο ίσως πολιτικές ομάδες να βρεθούν σε αντίθεση ε, στο ένα ή στο άλλο σημείο. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι θα πρέπει να συμβιβάσουμε και να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να βγάλουμε μια καλή έκθεση, όχι σαν έκθεση δική μου, σαν έκθεση όλης της ομάδας της Επιτροπής μας, διότι θεωρώ ότι πρέπει να εργούμε συλλογικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλαβράκο. Να σας υπενθυμίσω τις προθεσμίες. 7 Μαΐου το μεσημέρι. Το μεσημέρι. 7 Μαΐου το μεσημέρι είναι η προθεσμία. Τώρα, μία αλλαγή ακόμα πρέπει να κάνουμε, γιατί υπήρξε μία ε, παρεξήγηση. Απλώς να βάλουμε το σημείο 7 πριν από το σημείο 6. Εάν οι εισηγητές του 6 και του 7 συμφωνούν, θα πάμε στο 7 πριν από το 6, πολιετές σχέδιο για τον ε, Βαλτικό Σολομό και μετά θα περάσουμε στο σημείο 6. Σύμφωνοι. Ήδη τον Νοέμβριο είχε παρουσιαστεί το περιεχόμενο της πρότασης αυτής και τώρα βρισκόμαστε σε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Απλώς να λάβετε υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό έχει αλλάξει. Το Μάιο θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεση, τον Ιούνιο στην Επιτροπή μας και το Σεπτέμβριο, αν θέλει ο Θεός, στην Ολομέλεια. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκρόμπαρτσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολιτές σχέδιο για το απόθεμα Σολομού της Βαλτικής. Στόχος εδώ πέρα είναι να εγκρίνουμε ένα κανονισμό που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και αλληλευτική πτυχή του ζητήματος. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει βάση για την έκθεσή μας. Συνεπώς, προκειμένου να εργαστούμε σωστά, αρχίσαμε μία ευρεία διαβούλευση. Ήρθαμε σε επαφή με τους ίδιους τους αλείς, Ζητήσαμε να μάθουμε ποια είναι η άποψή τους, τι πιστεύουν για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους τοπικών κυβερνήσεων, καθώς επίσης και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, που και αυτοί με τη σειρά τους ενδιαφέρονται πολύ για το ζήτημα των πληθυσμών Σολομού. Μιλήσαμε επίσης με πολλούς ανθρώπους στη Φιλανδία και στη Σουηδία ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε ότι στις δύο αυτές χώρες έχουμε ποταμούς οι οποίοι έχουν πάρα πολλούς σολομούς. Μιλήσαμε επίσης και με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Και ήρθαμε σε επαφή επίσης και με πολλούς επιστήμονες. Τέλος, διοργανώσαμε μία συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε μία σύντομη ανταλλαγή απόψεων και σας έστειλα και μάλλον έστειλα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία σειρά από ερωτήσεις. Ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την συλλογή πληροφοριών για την εθνική νομοθεσία σε διάφορα κράτη-μέλη. Το πόρισμα λοιπόν όλης αυτής της διαβούλευσης ήταν ότι δεν έχουμε ακόμα αρκετές πληροφορίες, δεν υφίστανται αρκετά δεδομένα. Ακόμα μας λείπουν λοιπόν κάποιες σημαντικές πληροφορίες και ως εκ τούτου κινδυνεύουμε να χάσουμε τον στόχο μας. Όπως σας είπα, είναι να πετύχουμε την, την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στις τρεις αυτές πτυχές ε, του ζητήματος. Τώρα, παίρνοντας σε πιο τεχνικές λεπτομέρειες. Αναφερόμαστε το κυρίως σε αλία αναψυχής αεραστεχνική μάλλον αλία, στην, περιοχή της ε, Βαλτικής. Πρόκειται για ένα τύπο αλίας που δεν υπόκειται σε έλεγχο. Πολύ συχνά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τα απαραίτητα δεδομένα που να πορεύουν από τον έλεγχο. Ή πολλές φορές έχουμε και πλήρη απουσία τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ακόμα και στις ίδιες τις συμβάσεις που υπάρχουν. Πολύ συχνά μιλάμε για σκάφη αναψυχής ή για άλλα αλλιευτικά σκάφη, για άλλου είδους αλλιευτικές, άλλου είδους ε, αλλιευτικών μεθόδων. Δεν μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε σωστά αυτού του είδους την αλληλεία την αριστεχνική λοιπόν αυτή αλληλεία, όπου όμως όπως βλέπετε επηρεάζει πάρα πολύ τα αποθέματα Σολομού. Επίσης, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια λένε κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ΡΑΚ ουσιαστικά θέτουν ένα αμφιβόλο την ίδια τη βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ουσιαστικά δεν συμφωνούν με την ανάλυση που γίνεται για το πώς επηρεάζονται τα αποθέματα Σολομού από τις διάφορες μεθόδους αλίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με τα περιφερειακά γνωμοτικά συμβούλια, αλλά αυτή η συνεργασία θα είναι αρκετά δύσκολη. Ήδη έχουμε συναντήσει κάποιε δυσκολίε στην συνεργασία που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Επομένως, δεν έχουμε την απαραίτητη βάση για να δημιουργήσουμε μια στρατηγική συνεργασίας. Τα περιφερειακά γνωμοτικά συμβούλια προτείνουν διαφορετικές λύσεις προκειμένου να προστατεύσουμε το σολομό της Βαλτικής. Όσον αφορά τώρα την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, Το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε στη συζήτηση είναι το ακόλουθο, ή μάλλον τα ακόλουθα. Εραστεχνική αλία, αλία αναψυχής και μια ιδιαίτερα περιοριστική προσέγγιση σε αυτή τη μέθοδο αλίας που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Θα πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό, μια για πάντα, έτσι ώστε να μην έχουμε να το μετωπίσουμε στο μέλλον, όχι μόνο για τον σολομό της Βαλτικής, αλλά και για τα υπόλοιπα είδη. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η αναπραγωγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι στο άρθρο 5 λέγεται ότι η αναπαραγωγή θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του 75%. Εμείς θεωρούμε ότι το επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι το επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι υψηλότερο και εμείς προτείνουμε 80%. Τώρα, όσον αφορά τον επανεμπλουτισμό στο άρθρο 13 Εδώ πέρα προβλέπεται μία περίοδος 7 ετών. Μετά την περίοδο αυτή όμως, μετά τα 7 αυτά έτη, θα πρέπει να σταματήσει ο πανεμπλουτισμός και ουσιαστικά θα έχουμε φτάσει σε φυσιολογικά επίπεδα αναπαραγωγή στους ποταμούς. Όλοι μας λένε όμως ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι σωστή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μετά από 7 έτη θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε την όλη διαδικασία αναπαραγωγής. Εμείς προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση. μετά την πάροδο τριετίας, θα πρέπει να γίνει μία αναθεώρηση. Θα πρέπει να ελέγξουμε δηλαδή αν ε, η φυσική αναπαραγωγή του άγριου σολομού είναι βιώσιμη. Ενδεχομένω δηλαδή αυτή η επταετή περίοδο που προβλέπεται στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγική. Υπάρχουν ε, πολλές περιοχές στις οποίες έχει γίνει επαναπλουτισμός για 20-25 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τους ελέγχους, γνωρίζουμε ότι ε, δεν έχουμε την απαιτούμενη παρακολούθηση και εποπτεία της αεραστεχνικής αλίας. Ξέρουμε ότι όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν. και τα κράτη-μέλη δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα αυτό. Από την άλλη όμως, κάνουμε και την ακόλουθη πρόταση. Λέμε ότι όλα τα λευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα βιβλία, μερολογίο που θα πρέπει να καταγράφεται όλη αυτή η δραστηριότητα. Μπορούμε να έχουμε κάποια μικρά σκάφη, ακόμα και τριών-τεσσάρων μέτρων, στα οποία όμω ε, θα είναι ίσω ιδιαίτερα δύσκολο να έχουμε μερολόγιο. Στο άρθρο 20 λέγεται ότι το 10% του ε, συνόλου των αλλιευμάτων θα πρέπει να ελέγχεται. Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι πολύ ψηλότερο. Να μιλάμε δηλαδή για ένα 50%. 50% όλων των εκφορτώσεων. Το 50% όλων των εκφορτώσεων θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο στα πλαίσια του πολιετού σχεδίου. Τώρα, για ποιο λόγο θέλουμε εμεί κάτι τέτοιο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν να αξιολογούμε την κατάσταση. Και τέλος, ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ιδιαιτέρως είναι η επίπτωση που μπορούμε να έχουμε σε άλλα είδη, όπως η κομοράνοι ή οι φώκες. Θέλουμε να γνωρίζουμε, θέλουμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε είναι οι επιπτώσει από τη δραστηριότητα αυτών των ειδών όσον αφορά τα αποθέματα σολομού, γιατί προφανώ τα ίδια αυτά τρέφονται με σολομό. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν αξιόπιστες ε, πηγές ε, πληροφοριών που θα μας επέτρεπαν να αξιολογήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο στην περιοχή της Βαλτικής. Ξέρουμε όμως ότι ο αντίκτυπος αυτός είναι τεράστιος. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στις ε, τεράστιες καταστροφές που έχουμε στα αποθέματα Σολομού εξαιτίας των Κομοράνων. και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην νότιο περιοχή της Βαλτικής. Αυτά είχα να σας πω. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Βαλέντσα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να περάσω σε τρεις κέρδιες προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα, στο πολιτή σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει και την ε, αλία αναψυχής και στους ποταμούς και στις λίμνες. Γιατί προς το παρόν αναφέρεται μονάχα η ρύθμιση στη Βαλική και σε λεκάνες ε, γλυκού νερού. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε από εκεί την ε, βιοτεχνική και την αλία αναψυχής, ψυχαγωγική αλία. Βάσει των επιστημονικών στοιχείων, αυτή η μορφή αλίας είναι ένα σημαντικό τμήμα των ε, πηγών, των αιτίων θανάτου λόγω αλίας του Σολομού της Βαλτικής. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί αυτή η μορφή. Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένε χώρες η αλία αναψυχής καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της, ε, των πόρων Σολομού. Πάνω από 40% των εθνικών ποσοστώσεων καλύπτονται με αυτή τη μορφή. Επειδή δεν αντανακλάται όμως σε συλλογή στοιχείων αυτή η μορφή αλίας, υπάρχουν ελλείψεις πραγματικές στο σύστημα διαχείρισης των σολομικών πόρων. Επίσης το θέμα των μεταφερομένων ποσοστώσεων, των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων για τους ε, ποταμούς. Έχουμε κάποιες ε, αμφιβολίες για μια τέτοια μορφή διαχείρισης για τους ποταμούς. Το να έχουμε λοιπόν μια τέτοια διαδικασία στους ποταμούς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Οι θαλάσσιες περιοχές είναι οι κέρυες για την σχετική σταθερότητα. Στις ε, περιοχές των εσωτερικών υδατήρων πόρων βέβαια έχουμε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι αυτές που επικρατούν στις θάλασσες. Πρέπει να έχουμε συστήματα ειδικά για τις ε, ποτάμιες περιοχές, τις ποτάμιες λεκάνες ειδικά για τα κράτη-μέλη και που εμπλέκονται και επίσης για τις τρίτες χώρες που εμπλέκονται. Η προσέγγιση της Κομισιόν εδώ είναι καινοτόμα και διαφέρει από, από άλλους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τα χέλια και μιλάω για τον αρμόδιο κανονισμό που έξερε το 2007 οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να υπάρξει ανάκαμψη του χελικού πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα είδη. Επίσης, η αύξηση των αποθεμάτων δεν μπορούμε να περιμένουμε με φυσικά μέσα να υπάρξει αύξηση των αποθεμάτων. πρέπει ε, να βοηθήσουμε και εμείς αυτή τη φυσική διαδικασία. Γιατί αν αποτύχουμε στο εγχείρημα αυτό τώρα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανακάμψουν ποτέ αυτά τα αποθέματα. Η αρχική λύση για, την, ε, ε, για τον εμπλουτισμό στην αρχή περιλάμβανε μονάχα ορισμένες περιοχές που είχε, είχαν σολομό. Σε όλες τις περιοχές όμως που θα μπορούσε να συμβάλλει αυτό το εγχείρημα στην αναπαραγωγή, στην άγρια αναπαραγωγή του ποταμούς, ποταμίσιου Σολομού θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η διαδικασία. Και αυτή είναι φυσικά μια οδός η οποία θα πρέπει να αυξήσει την ανάπτυξη αυτού του είδους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρίστενσεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα πρόγραμμα διαχείρισης ε, του Σολομού της Βαλτικής και είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η κατάσταση των ε, αποθεμάτων ε, και θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την διαθεσιμότητά του και εμείς ε, συμμετείχαμε στην προπαρασκευαστική φάση για την έκθεση αυτή και γι' αυτό θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή. Ωστόσο θα ήθελα να σταθώ στις προτάσεις που υποβάλλουν οι πράσινοι. και που στην ουσία σημαίνουν ε, απόλυτη παγόρευση του, της αλληλείας του Σολομού. Νομίζω πως ε, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν πολύ δραστικό. Θα σήμαινε την άμεση πάυση οποιασδήποτε δραστηριότητας αλληλείας ε, του Σολομού. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ελέγχεται κάθε είδος αλληλεία συμπεριλαμβανομένου και αυτού, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ε, μεγάλου ποσοστού παράνομης αλληλεία ε, του Σολομού. Γι' αυτό και θα πρέπει τα μέτρα να είναι γενικά, να επιτρέπουν ελέγχους και να επιτρέπουν την κατάλληλη διαχείριση. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ανθρώπινων προδιαγραφών που καθορίζουν ε, την εγκατάσταση των πληθυσμών και των ηχθικών αποθεμάτων και στην περίπτωση του Σολομού. Αλλά πρέπει να προτείνουμε μέτρα τα οποία να είναι στοχευμένα και που θα επιτρέπουν να εξαλείφονται τα επικίνδυνα εμπόδια. Όσον αφορά τα 65 εκατοστά, που προτείνει η τροπολογία 311 και αυτό θεωρώ πως είναι πολύ δραστικό ως μέτρο όπως και η τροπολογία 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πάντως ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να έχουμε τελικό αποτέλεσμα θετικό. ο κύριος Κούν. Ο κύριος Βαλέντσα μίλησε ήδη εξ ονόματος της ομάδας μας και εγώ μπορώ να αποσύρω την αίτησή μου για χρόνο ομιλίας. Ευχαριστώ από την Κομισιόν. Κύριος Η κυρία Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μας έχει καλέσει. Ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια του εισηγητή. Δεν συμφωνώ απολύτως ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Φυσικά κάθε φορά πρέπει να δουλέψουμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν ε, συλλέγει δεδομένα για την ανασύσταση των αλλιευμάτων, ε, ωστόσο υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία τα οποία εκπονούν διάφορα επιστημονικά σώματα για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και που αφορούν το Σολομό. Ιδιαίτερα η Helcom συλλέγει στοιχεία για την ανασύσταση των ε, αποθεμάτων, στοιχεία τα οποία δεν συμπεριληφθήκαν στην αρχική μα πρόταση, διότι θεωρούσαμε πως ήταν βάρο για τα κράτη-μέλη το να διαχειριστούν την ανασύσταση ε, τι μάλλον τη συλλογή και τον έλεγχο των ε, δεδομένων για την ανασύσταση των στόκ. Ωστόσο, είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο και γνωρίζουμε πως η ανασύσταση των αλλιευμάτων είναι σημαντικό ε, στοιχείο για ορισμένα αλλιεύματα. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί στην έκθεση και σε κάθε ερώτηση που μπορεί να έχετε για διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρόμπατσερ, για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η ελπίδα μου είναι ότι θα μπορέσει να μας δοθεί αυτή η γνωμοδότηση το ταχύτερο δυνατό για το ελάχιστο μέγεθος. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό έχει αντιμετωπιστεί με κάπως περιοριστικό τρόπο. Με πάση περιπτώσει νομίζω θα είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Για τον Σολομό λοιπόν και την Πέστροφα έχει καθοριστεί ένα ελάχιστο μέγεθος αλλά ξέρουμε λόγω της βιολογίας των ε, ειδών αυτών ότι 65 εκατοστά για την Πέστροφα είναι πολύ, μεγάλος, ε, πολύ μεγάλο μέγεθος. Αυτά είναι σχετικά μικρόσωμα ψάρια. Τώρα για την Κομισιόν το θέμα της ε, αλίας αναψυχής για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς βασιζόμαστε στο γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει αρκετά στοιχεία για αυτή τη μορφή αλίας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να γυρίσουμε τώρα στο σημείο 6. Αλληλεία, ε, και μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής, ε, της αλληλευτικής ε, πολιτικής. Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στο παρελθόν, το Μάρτιο είχαμε μια νέα συνάντηση και τώρα έχουμε την τρίτη ευκαιρία και δίνω το λόγο στον κύριο Φιρέιρα για το θέμα αυτό, για να παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσή του. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση που έχετε ενώπιόν σας για την ε, μικρή αλληλεία και τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όπως θα διαπιστώσετε, στην ουσία περιλαμβάνει τις βασικές γραμμές που ε, είχατε δει στο έγγραφο εργασίας που ήδη συζητήσαμε δύο φορές. Σε αυτές τις συζητήσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, και πικοδομητικές, ακούσαμε συμβολές διαφόρων ε, συναδέλφων και ακούσαμε, είδαμε και τις γνωμοδοτήσεις της Περιφερειακής Επιτροπής και της Επιτροπής των Γυναικών που ήταν πολύ χρήσιμες συμβολές για αυτή τη συζήτηση και για αυτή την έκθεση. Τελικά ε, είναι δύσκολο να συμπυκνώσει κανείς 6.000 χαρακτήρες όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα εργασία και στις ε, συμβολές των συναδέλφων και των άλλων επιτροπών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα σημεία τα οποία ήταν τα πιο σημαντικά συμπεριλήφθησαν εδώ. Βέβαια, μπορούμε πάντοτε σε αυτή τη φάση των τροπολογιών να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία, κάποια σημεία και να προσθέσουμε ίσως. που λόγω αυτού του ορίου έμειναν εκτός. Μπορούμε τώρα λοιπόν να τα προσθέσουμε ε, με έτσι των τροπολογιών. Πολύ σύντομα που τα θέματα που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά είναι καταρχήν η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας ε, της μικρής αλ... παράκτης ε, και η λογική συνέπεια που κάτι τέτοιο πρέπει να έχει στη διαφορετική αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης αλληλείας. Πρέπει να προβλεφθούν ε, καθεστώτα και μοντέλα διαχείρισης που θα λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες αυτού του, αυτού του είδους της αλληλείας. Έπειτα χρειάζεται μια δεν χρειάζεται μάλλον μια, ένας ορισμός περιοριστικός στις μικρές αλληλίες Και εδώ προσπαθώ να δείξω ορισμένες διαστάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν ορίζουμε την έννοια της μικρής αλληλίες. Διαστάσεις που ξεπερνούν το αυστηρό κριτήριο των διαστάσεων των σκαφών. Έχουμε και το θέμα που σχετίζεται με το θέμα της εγκύτητας σε αντίθεση με την κεντρικό χαρακτήρα της αλίας όπως έχει ε, σχηματιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και αν συνεχιστεί αυτή και εγκριθεί η πρόταση της Κομισιόν έτσι όπως ε, προτείνεται και μέχρι στιγμής, θα συνεχιστεί αυτή η κεντρική εικόνα και αυτή η τάση συγκέντρωσης που βέβαια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω του ότι δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις διάφορες πραγματικότητες επειδή υπάρχει ε, επίσης ε, η διαφορά των τομέων που δεν συμμετείχε στην εκπόνηση αυτής της μεταρρύθμισης και λόγω της διαφοράς στις στα διάφορα λιεύματα και στα διά, στους διάφορους στόλους ε, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάτι ακόμα είναι η απόρριψη απέναντι σε αυτή τη μεγάλη διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει την αλληλεία στα κράτη-μέλη, η επιβολή ενός ενιαίου μοντέλου, μοναδικού μοντέλου διαχείρισης είναι ακατάλληλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης, ε, για την λήψη μέτρων προσαρμοσμένων στη δική τους πραγματικότητα. Και στην περίπτωση των δικαιωμάτων, των δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαλέγουν και να μπορούν να αποφασίσουν ποια κομμάτια του στόλου εμπίπτουν ή όχι, μάλλον διέπονται ή όχι από αυτό το σύστημα. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και εδώ είναι μια πτυχή που αναφέρθηκε στην έκθεση. Πέρα από την όγκο του στόλου, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη και η ποιότητα του στόλου. Δεν αρκεί να προωθήσουμε μια μείωση γενική των, του στόλου για, με βάση μάλλον κριτήρια της αγοράς αποκλειστικά, αυτό προτείνει η Κομισιόν να προωθήσουμε λοιπόν αυτή τη μείωση της, των δυνατοτήτων μέσω της λειτουργίας αυτής της αγοράς αυτών των, των δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να σημαίνει απλά και μόνο μια συγκέντρωση της προσπάθειας της αλληλείας για τους ε, φορείς που είναι πιο ανταγωνιστικοί αποκλειστικά από οικονομικής άποψης. Μπορεί δηλαδή να καταργήσουμε διάφορα σκάφη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η πίεση στα αποθέματα θα μειωθεί, γιατί αυτά που θα μείνουν μπορεί να συνεχίσουν την ίδια προσπάθεια και παραπάνω. Και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την ποσότητα, τον όγκο του στόλου, αλλά και την ποιότητα και να καταβάλουμε μια προσπάθεια ώστε να κυριαρχήσει στο μέλλον να κυριαρχήσει στο μέλλον στη σύσταση των στόλων των κρατών μελών να κυριαρχήσουν περισσότερο εκείνα τα κομμάτια τα οποία είναι πιο βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και από άποψη οικονομική και κοινωνική. Και αυτό δεν είναι εγγυημένο με το σύστημα των δικαιωμάτων που προτείνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα παραμείνει θα είναι μόνο εκείνα τα κομμάτια, τα πιο ανταγωνιστικά από οικονομική άποψη και όχι αυτά που είναι πιο βιώσιμα από υπερβαλλοντική ή κοινωνική άποψη. Και αυτό όταν μιλάμε για μικρή αλληλεία έχει τεράστια σημασία και εγώ επιμένω για την, ότι οι δικλείδες ασφαλείας που προβλέπει η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, δεν αρκούν για την επιβίωση αυτής της μικρής αλληλείας και μπορούμε να δούμε τη ζημιά που έχει προκληθεί στις χώρες όπου το σύστημα αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί. Κάτι ακόμα σε σχέση με την εκπόνηση ενός κοινοτικού προγράμματος για τη στήριξη της μικρής αλίας που ε, συγκεντρώνει διάφορα υπάρχοντα μέσα, το μελλοντικό Ταμείο ε, Αλίας και άλλα μέσα της πολιτικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, όλα αυτά διαρθώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίξουν τον τομέα της μικρής αλίας μέσω ενός κοινοτικού προγράμματος στήριξης στη μικρή αλία. δίνεται η εγγύηση για ένα μίνιμουμ ποσό του μελλοντικού ταμείου αλληλείας σε αυτά τα τμήματα της μικρής αλληλείας, τους φορείς της μικρής αλληλείας, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης από τον Ταμείο Αλίες σε σχέση με την κοινή οργάνωση της αγοράς για τα προϊόντα ε, αλίες και υδατοκαλλιέργειας θεωρούμε ότι η ΚΟΑ θα πρέπει να αυξήσει τη συμβολή της ώστε να εγγυηθεί ένα δίκαιο εισόδημα στον τομέα της μικρής αλίας. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η συμβολή της ε, για τη σταθερότητα των αγορών αλλά και για τη βελτίωση της ε, ε, πορεία των προϊόντων αυτών. Η αξιολόγηση που κάνουμε είναι ότι από όσο γνωρίζουμε από την πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή την αποσύνθεση των μέσων ρύθμισης της αγοράς δεν θα είναι ωφέλιμο για τη μικρή αλληλεία. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν αυτά τα μέσα σταθεροποίησης της αγοράς για να συντηρηθεί η μικρή αλληλεία, γιατί είναι ένας από τους πυλώνες της κοινή οργάνωσης αγοράς και θα μπορεί έτσι να έχει ένα δίκαιο εισόδημα όποιο περιμένει να ζήσει από αυτή τη δραστηριότητα. Στην... Και ολοκληρώνω. Στην έκθεση υποστηρίζουμε μηχανισμούς ε, επίγουσας ανάγκης, δηλαδή μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις επίγουσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρή αλληλεία είναι πιο ευάλωτη από ότι άλλοι είδους αλληλείες σε εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή για παράδειγμα σε μια ξαφνική αύξηση του κόστους παραγωγής, όπως ας πούμε των καυσίμων, είτε λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε πιστώσεις. Η αντοχή λοιπόν της μικρής αλίας είναι πολύ μικρότερη σε όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες και σε σχέση και με τη συζήτηση που έγινε πριν για την έκθεση του συναδέλφου Σαλα, ε, Σαλαβράκου. Ορισμένα, ορισμένες από αυτές τις μικρές αλίες μπορεί άμεσα να επηρεαστούν από την αύξηση των καυσίμων. Η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά θα αντιδράσει. Η μικρή αλία λιγότερο μπορεί να αντισταθεί απέναντι σε αυτές τις ε, απότομες διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής. Θα πρέπει αυτό να είναι το σημείο εκκίνηση για να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτού του είδου αλληλεία, αν θέλουμε να το διατηρήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν δηλαδή μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και αυτές ε, οι προτάσεις περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Τέλο η περάσπιση μιας αρχής και μάλιστα η διεύρυνση της ε, περιοχής αποκλειστικής ζώνης που είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη. Όλοι θεωρούν ότι είναι θετική η ζώνη αυτή, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην θεσπιστεί λοιπόν ω μόνιμη αρχή, εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα και να διευρυνθεί κάπω κιόλα. Εμείς θα θέλαμε αυτή η διεύρυνση να πρέπει να γίνει σύμφωνα και με την υφαλοκρηπίδα, να επεκταθεί ως τα 12 μίλια. Υπάρχουν ευαίσθητες περιοχές ε, αλληλείας και η ζώνη αυτή κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να επεκταθεί και να καλύπτει το σύνολο της αποκλειστικής οικονομικής ε, ζώνης ή αλλιώς να επεκταθεί από τα 100 στα 200 μίλια. Θα περιμένω λοιπόν τις παρατηρήσεις και των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Πέντε ομιλητέ θέλουν να λάβουν το λόγο. Έξι. Δύο λεπτά σας παρακαλώ. Επτά. Δύο λεπτά. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα, βγάλουμε ακριβή. Κύριε Φράγα. Ευχαριστώ. Προσπαθήσω να παραμείνω μέσα στα δύο λεπτά που μου δίνετε. Πρώτα απ' όλα, για την έκθεση του εισηγητή, εγώ θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του να έχουμε ένα νέο ορισμό παράκτιας αλίας που να περιλαμβάνεται στην κοινή αλλιευτική πολιτική είναι πάρα πολλά τα κριτήρια που υπάρχουν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα διαλέξουμε μόνο ένα και θα αγνοήσουμε τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα νέο τρόπο να καθορίσουμε τι σημαίνει παράκτια αλία, που να είναι πιο πλήρη ορισμό από αυτόν που έχουμε. Δεύτερον, για τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Η κύρια επιφύλαξή σας για το θέμα αυτό δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι η πρόταση της Κομισιόν επιτρέπει η παράκτια αλία να εξαιρεθεί από την χρήση των μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχει νόημα η επίκρισή σας γιατί κάνετε επίκριση σε κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσετε διότι θα παρέμβει επικουρικότητα για το θέμα αυτό. Μου φαίνεται ότι είναι υπερβολικό λοιπόν αυτό που λέτε για τις μεταφερόμενες ποσοστώσεις. Το ότι η κρίση θίγει κυρίως την παράκτια αλία, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει η κρίση ε, πλήττει κυρίως τις μορφές αλίας που καταναλώνουν περισσότερο πετρέλαιο στην πράξη. Για την αλλιευτική ικανότητα που αναφέρεται στο σημείο 8, πιστεύω ότι εκεί η παράκτεια και βιοτεχνική αλληλεία πρέπει και αυτή να προσαρμοστεί στους ε, αλλιευτικούς πόρους. Δεν είναι σωστό να πούμε ότι για την βιοτεχνική αλία και την παράκτη αλία δεν υπάρχει πρόβλημα υπεραλίευσης. Τονίζω λοιπόν ότι δράτη, ε, ότι μάλλον δρά η παράκτη και η βιοτεχνική αλία στα πιο ευαίσθητα από όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα, επομένως θα πρέπει και εκεί να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης της ε, αλευτικής ικανότητος, εάν και πιστεύω ότι πολύ συχνά ισχύει αυτό, είναι απαραίτητο. Και κλείνω. Και κλείνω διότι έχω περάσει και τα δυο μου λεφτά. Η ελευθερία πρόσβασης, αυτή είναι μια βασική αρχή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει το όριο των 12 μιλίων για καλύτερη προστασία της παράκτειας Αλίες Λέτε ότι αυτό θα πρέπει να φτάνει στα 200 μίλια για τις υπερπεριφερειακές περιοχές, αλλά αυτό δεν αφορά την βιοταχνική αλία. Οποιαδήποτε εξαίρεση θα πρέπει να την χάνει ε, αιτιολόγησης και δεν νομίζω ότι αυτοί που αλλιεύουν 200 μίλια μακριά από τη βάση τους βρίσκονται στα πλαίσια της βιοτεχνικής αλίας. Ο κύριος Μπεσέτ. συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να επαναλάβω κάποιες γενικές αρχές, γιατί δεν έχουμε χρόνο να περάσουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η έκθεση του κυρίου Φερέιρα θεωρούμε ότι κινείται σε θετικό δρόμο θα καταθέσουμε βέβαια και τροπολογίες προκειμένου να εμπλουτίσουμε το κείμενο σε διάφορα σημεία. Βλέπουμε σε μια πρώτη φάση ότι προσπαθεί να καταλήξει σε έναν νέο ορισμό της παράκτειας παραδοσιακής βιοτεχνικής αλίας και ότι προσπαθεί να διευρύνει τον ορισμό αυτό προκειμένου να καλύψει περισσότερο τη μορφή αυτή αλίας, να συμπεριληφθούν δηλαδή και άλλα κριτήρια πέρα από αυτά τα οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Φράγκα κάνει και αυτή μια πρόταση ορισμού σε ένα άλλο όμως πλαίσιο. Πολύ καλά. Πιστεύω όμως εγώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο στην προσπάθεια αυτή να ξέρουμε εξ αρχής για το τι μιλάμε. Δεύτερον, η έκθεση του κυρίου Φερέιρα προσελκύει την προσοχή μας σε μία μορφή δραστηριότητας, δηλαδή στην παράκτη αλία, την αλία μικρής κλίμακας, η οποία δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας και ουσιαστικά δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας από τις άλλες μορφές αλίας και καταναλώνει και λιγότερους πόρους. Κυρία Φράκα, νομίζω ότι διαφωνούμε εδώ πέρα. Επί της ουσίας όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της αλίας μικρής κλίμακας και ότι θα πρέπει αυτή να συμπεριληφθεί στην νέα κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να προβλέψουμε εδώ πέρα ένα καθεστώς παρέκκλησης, εξαίρεσης για αυτή την αλλία. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια μορφή αλίας η οποία τελικά δεν θα υπάγεται στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της ε, νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής προκειμένου να προωθηθούν ακριβώς αυτά τα οποία λέτε και εσείς στην εκθεσή σας. Διατήρηση συντήρηση των πόρων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Κύριο briefly, um, Κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, περισσότερες θέσεις εργασίας στην παράκτη αλληλεία, ναι, βεβαίω. Αλλά όλα αυτά με ελάχιστο κόστος προς το περιβάλλον κατανοώ ότι όπως λέει η κυρία Φράγκα δεν ισχύει αυτό πάντα, ένα 12 μέτρο πλοίο μπορεί να πιάσει πολλά ψάρια. Πολλά ψάρια. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλη η αλία αναψυχής είναι φιλική προ το περιβάλλον. Τρία σημεία. Ίσως ξαναλέω κάτι για τι μεταβάσιμες ποσοστώσει που το έχω πει 40 φορέ. Το έγγραφο εργασία όμω λέει ότι το, η πρόταση τη Κομισιόν υποβάλει την πρόσβαση στους, ε, στους αλληλευτικούς πόρους με ένα μονάχα σύστημα. <coughs> Δεν είναι το ίδιο σύστημα με τα ITQ της ε, ατομικές ποσοστώσεις. Μπορεί κανείς σε εθνικό επίπεδο να καθορίσει τις ποσοστώσεις όπως θέλει και ένα από αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι η προστασία της μικρής αλλίας και των παρακτήων κοινοτήτων. Υπάρχει τώρα και ένα θέμα κονδυλίων. Ναι, επικαλύπτεται με κάποιους από τους στόχους της Κομισιόν για να υποστηριχθούν οι παράκτιες κοινότητε και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. Αλλά αν δώσετε σε ένα τμήμα μοναχα των αλλιέων κάποια χρήματα, κάποιοι άλλοι θα πάρουν λιγότερα λεφτά. Αυτό εντάξει, αλλά εξαρτάται από το ποια είναι η πρότασή σα. Δεν κατάλαβα το επιχείρημα των αζωρών έχουν 100 μίλια και θέλετε να πάτε στα 200 μίλια. Πολύ θάλασσα, πολύ ψάρι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν ξέρω αν το επιχείρημά σας δικαιολογεί αυτό το οποίο λέτε. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέιβις. Ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Μπορώ να μιλήσω ειδικά. Είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετέχω και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου και εκεί συζητούμε το θέμα αυτό. Πήρα λοιπόν στην Επιτροπή αυτή τον λόγο και αναφέρθηκα στην ε, υδατοκαλλιέργεια, στις, στους μηχανισμούς υδατοκαλλιέργειας που έχουμε στη Βόρεια Ευρώπη, που είναι μορφές ε, υδατοκαλλιέργειες πάρα πολύ σημαντικές και δημιουργούν και πολλές θέσεις ε, εργασίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υδατοκαλλιέργειες μικρής κλίμακας. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις υδατοκαλλιέργειες αυτές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πολύ στην Βόρεια Ευρώπη και θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα αυτό. Φέρει και αυτό ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Η κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ την κυρία Κρέσπο για τις νέες της ευθύνες και θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν για το σημείο 11 όπου μιλάει ο εισηγητής για την υποστήριξη σε πρακτικές ε, οι οποίες είναι βιώσιμες σε ό,τι αφορά την συλλογή των οστρακοειδών. Στα ισπανικά τώρα λέγεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα θέμα ε, γλωσσικό στη μετάφραση. Πρόκειται για συλλογή οστρακοειδών αλλά και εκτροφή τους, γιατί και αυτό γίνεται με τρόπο ο οποίος είναι βιώσιμος και αηφόρος στη Γαλλικία έχουμε 17.000 θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Επίσης το σημείο 14 εσείς υποστηρίζετε τη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως είναι φυσικές καταστροφές κτλ. Θα πρέπει να έχουμε και μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για περίπτωση ρήπανσης με πετρέλαιο, <clears throat> για μολυσμένα νερά, σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε παραδείγματος χάρη στην ε, Γαλλικία, η οστρακο παραγωγή εκεί πέρα πρέπει να, να έχουν προστασία από ανθρώπινες από ανθρωπογενείς καταστροφές οι οποίες τους δημιουργούν προβλήματα. Όλες αυτές λοιπόν οι κοινωνικές πτυχές που μπορούν να προκύψουν από καταστροφές ανθρωπογενείς όπως είναι τα ατυχήματα πετρελαιοφόρων κτλ. πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μιράντα. Κύριο κύριος Σάντσεφ Πρεσέδο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ σύντομα να πω ότι υπάρχουν ορισμένε πτύχες που έχει σωστή αντιμετώπιση σε αυτά ο κύριος Φεραίρα και μπορούμε να ενισχύσουμε λιγάκι τις κατευθύνσεις αυτές, καταρχήν σε ό,τι αφορά τον ε, ορισμό, πότε ψαρεύει κανείς, ε, πού ψαρεύει, τι ψαρεύει, με τι αλλιευτικά, ε, αλλιευτικό εξοπλισμό και τεχνική. Μπορούμε λοιπόν εκεί να έχουμε και μια μεγαλύτερη ενίσχυση και να τονίσουμε και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της αλίας και όχι μονάχα το γεγονός ότι προστατεύει το περιβάλλον. Να τονίσουμε λοιπόν το θέμα της ε, πολυμορφίας δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την αλία. Και η βιοτεχνική αλληλεία και η παράκτια αλληλεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παράλληλα με τη μικρή κλίμακος η χθιοκαλλιέργεια που γίνεται παραδοσιακά στις περιοχές αυτές και σε σχέση με την εμπορία θα πρέπει να τονίσουμε την καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή για τα νοπά προϊόντα και να εξασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των ίδιων των αλλιέων στα συστήματα διαχείρισης. Ο κ. Μιλάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με την θέση του Φερέιρα, αλλά και με κάποια πράγματα που είπε συνάδελφο ε, Φράγκα. Δεν είναι όλοι οι αλλοί οι ίδια. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και με τον Ντέιβις. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές ε, που μπορεί να βλάψουν ιδιαίτερα το περιβάλλον, ιδιαίτερα αυτό που είναι το κοντινό στις ακτές, το 12 με 100 μίλια. Πολλές φορές ένα μικρό σκαφάκι που αλλιεύει παράκτια πολύ συχνά προκαλεί ζημιές πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μεγάλα σκάβη που αλλιεύουν πολύ πιο μακριά και γι' αυτό και ο ορισμός είναι πολύ σημαντικός και θέλω να ζητήσω από το Φερέιρα να το σκεφτεί και να διευκρινίσει καλύτερα αυτή την ε, πτυχή. Μια άλλη ερώτηση. Για πολλές χώρες η προσπάθεια της αλληλείας σχετίζεται και βασίζεται και στην μικρή αλληλεία και πολλές φορές προκαλεί παραλογισμούς. Δηλαδή, να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και θα κλείσω με αυτό που υπάρχει στην Ιταλία, αλλά νομίζω σε ολόκληρη τη Μεσόγειο η αλληλευτική προσπάθεια ορίζεται με περισσότερες δεσμεύσεις. Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι μικροί τοπικοί αλληλείες που έχουν ακόμα κινητήρες που ίσως να υιοθετούν το σύστημα της αλληλείας με σταθερό δίχτυ που δεν μπορεί να είναι πιο μακρύ από 4 χιλιόμετρα, όπως δεσμεύεται από την Αλία για τη Μεσόγειο, και ταυτόχρονα δεν μπορούν να έχουν ε, μοτέρ μεγαλύτερο από αυτό που ήδη υπάρχουν. Και υπάρχει ένα μεγάλο στόλος αλιών που αλλιεύει με ε, μοτέρ 5 ύπων, δηλαδή με πολύ άσχημες συνθήκες και ασφάλειας, γιατί ο κανονισμός για τη Μεσόγειο έχει υποχρεώσει να αλλιεύουν πέρα από τα 12 μίλια. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε δύο πράγματα. Ορισμός της μικρής παράκτης αλίας και ορισμός της αλληλευτικής προσπάθειας που συμβάλλει που, μάλλον που περιλαμβάνεται στην εθνική αλληλευτική προσπάθεια. Κατά τα λοιπά συμφωνώ απόλυτα και για το γεγονός ε, ότι το ΦΕΜΠ θα πρέπει να δημιουργήσει και ίσως και εις βάρος άλλων μια γραμμή βοήθειας για τη μικρή παράλια, ε, παράκτια αλληλεία. από τη στιγμή που αποδεχόμαστε πως αυτή συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν θέτει σε κίνδυνο την ε, δυνητική ανασύσταση των ε, αποθεμάτων. Όσο πιο αυστηρός όμως είναι ο κανονισμός, ο ορισμός με συγχωρείτε της μικρής αλλιευτικής ε, αλίας, τόσο πιο πετυχημένες θα είναι οι δράσεις ε, της αρρωγής που θα προβλέψουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μιλάνα. Κυρία... Ευχαριστώ κυρία Λοβέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπε και ο συνάδελφος από τους Πρασίνους, ο κύριος Μπεσέ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η αλία μικρή κλίμακα χρειάζεται ένα τόσο ξεχωριστό κανονισμό. Ουσιαστικά φαίνεται να την αποκλείουμε από την κοινή αλληλευτική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να πούμε ότι ορισμένες αρμοδιότητες μπορούν να παραχωρηθούν στα κράτη-μέλη, να διευθετηθούν δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, πιστώσεις όσον αφορά την αλία μικρής κλίμακας ή επιπρόσθετες ποσοστώσεις για φωτίδου στην αλία. Το πιο σημαντικό πάντως είναι η αλία μικρής κλίμακας να είναι βιώσιμη, να προστατεύει το περιβάλλον και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι πιο σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης. Στο σημείο 11 της έκθεσής σας, τουλάχιστον στην αγγλική εκδοχή της έκθεσης, λέγεται ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα για τον εξυγχρονισμό, την ανανέωση. Στο σουηδικό κείμενο λέγεται Renovation και Modernization. Αναφέρεστε εδώ πέρα σε νέα σκάφη, για παράδειγμα. Δεν νομίζω θα πρέπει χρηματοδοτικά εμείς να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, αν σε αυτό αναφέρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν, Κομισιόν έχει κ. Σας ευχαριστώ. Ναι, προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα χρηματοδοτούσε ποτέ την ανανέωση ανακαίνιση σκαφών. Δεν θα ασχοληθώ με το ζήτημα του ορισμού. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει, σας το έχουμε εξηγήσει. Εσείς θα κάνετε τη δική σας συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Είναι σαφώς πάντως από την πρότασή μας ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μη διαφοροποιημένο καθεστώς. Αντίθετα θέλουμε διαφοροποιημένο καθεστώς για τους μεγάλους και τους μικρούς στόλους αυτό γίνεται σε κάποιες πτυχές της πολιτικής και ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των στόλων και τα TFCs, τις μεταβάσιμες παραχωρήσεις. Όπως είπε η κυρία Φράγκα, προβλέπεται να μην συμμετέχει η αλία μικρής κλίμακας ή μικρής στόλη στα TFCs. Και επίση, και αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται βέβαια στην πρόταση αυτή, προβλέπονται σαφεί εξαιρέσει από το καθεστώ ελέγχου γιατί είχε θεωρηθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό και θα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό γραφειοκρατικό άχθος για τους μικρούς στόλους. Και τέλος, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει απαραίτητη διαφοροποίηση ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους στόλους. Για πρώτη φορά όμως, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο το μέγεθος του, των σκαφών του μικρού στόλου ανά κράτος μέλος και ότι αυτό ουσιαστικά θα πειράσει και το ζήτημα της χρηματοδότησης. Δεν έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό άρθρο, αλλά θα προκύψει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται όμως στην έκθεση και πρέπει να το αναφέρω. Επιμείναμε πάρα πολύ και υπόθηκε γι' αυτό σήμερα, στο ότι θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικέ διατήρηση, συντήρηση και θα πρέπει να ισχύουν για οποιοδήποτε σκάφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το μέγεθό του, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τη αλληλεία στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτό που θέλουμε να συντηρήσουμε, διατηρήσουμε είναι τα αποθέματα βέβαια και όχι ο στόχο. Θα πρέπει λοιπόν διασυνοριακά να ισχύουν τα ίδια μέτρα. Και δύο ακόμα παρατηρήσει. εκεί όπου ο εισηγητής αναφέρεται στις ε, τοπικές, ε, στα τοπικά μέτρα διαχείρισης, εμείς αντιπροτείνουμε τα όσα λέμε για την περιφερειοποίηση και τα όσα λέμε για τις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να έχουμε καλύτερα μέτρα διαχείριση σε τοπικό επίπεδο και μέσω της περιφερειοποίησης κάποιες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν από τις ίδιες τις παράκτιες ε, περιφέρειες και περιοχές. Στα πλαίσια επίσης της κοινή οργάνωσης αγοράς, μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο των οργανώσεων παραγωγών πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εντοπισμένη, ε, τοπική μάλλον, ε, διαχείριση της αλίας και σε υπεράσπιση κατά αυτόν τον τρόπο των τοπικών μικρών στόλων. Βέβαια, στην κοινή οργάνωση αγορά ή μέσω τη κοινή οργάνωση αγορά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπέ εισόδημα για όλου του αλληλεί. Δεν μπορεί να είναι στόχο αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, στρατηγική της αγοράς, τη στρατηγική παραγωγής και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε και καλύτερα εισοδήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο έκθεσης και προσβλέπουμε στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ <clears throat> κύριε Φεραίρα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στη συζήτηση κάποια σχόλια για συγκεκριμένα θέματα. Τι είναι ο σωστός ορισμός της μικρής αλίας. Κατανοώ την ανάγκη να έχουμε ένα σαφή ορισμό, όπως το ανέφερε η κυρία Φράγκα. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να υπάρχει προτιμησιακή πρόσβαση στα ταμεία αλίας η μικρή και βιοτεχνική αλία, θα πρέπει να έχουμε ένα αντικειμενικό ορισμό του ποια είναι αυτή η μορφή αλίας που θα τύχει προνομιακής μεταχείρισης. Και στην ε, τελευταία μας συνεδρίαση η κυρία Φράγκα έκανε μια πάρα πολύ χρήσιμη συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Μίλησε για την ε, διάρκεια της αλληλευτικής δραστηριότητας ως μια βάση για, την, ε, για τον καθορισμό της ε, αλίες. Επίσης, συμφωνώ με την ιδέα η παράκτη αλία, η μικρή αλία, όπως και οι άλλες μορφές αλίες να προσαρμοστούν στους διαθέσιμους πόρους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και η κυρία Λόβιν επίσης το θέμα αυτό. <clears throat> Δεν υπάρχει κάποιο σημείο στην έκθεσή μου που να προτείνει η μικρή, μικρής κλίμακος αλία να μην υπόκειται στους κανόνες προστασίας και διατήρησης των αλληλευτικών πόρων. Πουθενά δεν λέω κάτι τέτοιο. Να αφήσουμε απ' έξω από τους κανόνες την μικρή κλίμακος Αυτό το οποίο διεκδικώ στην έκθεση αυτή είναι το νομοθετικό πλαίσιο να μην, είναι, να μην αποβεί σε βάρος της μικρής αλίας και στο βαθμό του δυνατού να κάνει θετική διάκριση υπέρ της. Γιατί ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες αυτού του, του, του τομέα και την ανάγκη να τον προστατεύσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να συνάδει με τη μελλοντική διατήρηση αυτού του τομέα και να μην οδηγήσει στον εξαθαναποδισμό του τομέα αυτού. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθώ εγώ να επιτύχω είναι το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο να είναι συμβατό όχι μόνο με τη διατήρηση αλλά και με την ενίσχυση του τομέα αυτού και την επίλυση πολλών από τα προβλήματα αυτού του τομέα. Δεν θέλω να τον αφήσω έξω από τους γενικούς κανόνες. Κάτι άλλο τώρα. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να το επιτύσσουμε αυτό και αυτό καταγράφεται στο σημείο 6 της έκθεσης το τι σημαίνει μια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο εγγύη εγκύτητος. Να σταματήσουμε λοιπόν να έχουμε μια κεντρική διαχείριση η οποία είναι μακριά από την πραγματικότητα και που περιλαμβάνει κατευθύνσεις οι οποίες δεν γίνονται κατανοητές από τους αλληλείς και δεν εφαρμόζονται στις συγκεκριμένε πραγματικότητες κάθε περιοχής και που ακόμα και με μεγαλύτερες δυνατότητες και πόρους ελέγχου δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μια τέτοια ρύθμιση και πολλές φορές έχει και αντιπαραγωγικό χαρακτήρα. Η αποκέντρωση λοιπόν της διαχείρισης είναι μια αναγκαιότητα. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ανεπαρκής η πρόταση περιφερικοποίησης της ε, Επιτροπής. Δεν ανταποκρίνεται στην κατεπίγουσα ανάγκη να υπάρξει διαχείριση σε επίπεδο εγκύτητο. Στο σημείο 6 λοιπόν προσπαθώ να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διαχείριση σε επίπεδο εγκύτητο. Είπε η κυρία Φράγα ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον αντίκτυπο που έχει η μικρής κλίμακος και βιοτεχνική αλία στους θαλάσσιους πόρους. Δεν λέω ποτέ ότι δεν έχει καμία επίπτωση, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Φράγκα. Αλλά επανερχόμαστε σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε λιγάκι καλύτερα ποια είναι η πραγματικότητα αυτού του τομέα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της μεταρρύθμισης είναι ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε μία πραγματικότητα η οποία ακόμα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό άγνωστη σε εμάς. Το λέει η Κομισιόν, λέει δεν έχουμε ακόμα τις μελέτες που ήδη από πολύ καιρό θα πρέπει να είχαμε σε σχέση με την υπερβολική αλίευση, του τομεί που υπάρχει υπερβολική αλίευση, σε ποια κρατημέλη, σε ποια τμήματα του στόλου, σε ποια αλλιευτικά είδη κτλ. Άμα θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε μια πραγματικότητα που δεν τη γνωρίζουμε καλά, ο κίνδυνος να κάνουμε λάθος είναι πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό θα πρέπει πάνω απ' όλα να βελτιώσουμε τη γνώση των ε, Τη κατάσταση των αλληλευτικών πόρων και σε σχέση με τη μικρή κλιμακοσαλία και την επίπτωσή τη στους πόρου. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για ορισμένου τομεί τη παράκτεια αλεία, για ορισμένα κράτη-μέλη, για ορισμένα είδη υπάρχει πράγματι υπερβολική ικανότητα, αν είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια τροποποίηση στου ε, πόρου σε αυτό το τομέα, εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μείνει απ' έξω η μικρή μικρή κλιμακοσαλία. Εκεί που μπορεί να έχω διαφορά μαζί σα είναι το πώ θα γίνει αυτή η προσαρμογή. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε. Η μία είναι η άποψη τη Κομισιόν. Η αγορά θα αποφασίσει και τέρμα. Δηλαδή είναι η πιο ανταγωνιστική από οικονομική άποψη οι οποίοι θα επιβιώσουν. η άλλη αντίο. Εγώ αντίθετα έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ότι δεν είναι μονάχα η αγορά η οποία πρέπει να λύσει όλα τα προβλήματα και υποχρεωτικά οπω λέει η Κομισιόν. Θα πρέπει να λαβουμε υπόψη και άλλα κριτήρια κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ανάγκη διατήρησης ορισμένων μορφών αλίας, με τα θέματα απασχόλησης, με τις σχέσεις απασχόλησης με ορισμένες μορφές αλίας, δηλαδή με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια αηφορίας και όχι μονάχα με το γνώμονα της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Και γι' αυτό σας λέω ότι η μείωση της ε, ικανότητας αλίας στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει δεν θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και υποχρεωτικά μέσω μηχανισμών αγοράς. Μπορούμε να έχουμε ένα πιο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αποφασίζεται όταν βλέπουμε, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει υπερβολική ικανότητα ότι ένα τομέα θα πρέπει να υποστεί τροποποίησεις χωρίς να είναι κατά μόνο με το μηχανισμό των μεταβιβασίμων ποσοστώσεων. Και εδώ δεν κάνω κάποια ε, διάκριση μεταξύ των ατομικών ποσοστώσεων και των μεταβιβάσιμων γενικά ποσοστώσεων. Ξέρουμε ότι υπήρξε αυτή η ανάγκη να αλλάξουμε το σύστημα έναντι των προηγούμενο που είχε αντιμετωπίσει πολλές ε, αντιδράσεις, αλλά για μένα δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική διαφορά μεταξύ των συστημάτων. Για τα 200 μίλια. Γιατί σε υπερπεριφερειακές περιοχές Μιλάω για 200 μίλια. Η κυρία Φράγκα, όχι ο κύριος Ντέιβις, ήταν μαζί μας στην αντιπροσωπεία που πήγαμε στις Αζόρες και άκουσε πολλές φορές από τα χείλη πάρα πολλών συνομιλητών ποιος είναι ο λόγος για να υπάρξει αυτή η διεύρυνση στα 200 μίλια. Σε περιοχές μεταξύ 100 και 200 μιλίων λειτουργούν στόλοι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στις τοπικές κοινότητες, αλλά δεν είναι εύκολο να τους εντάξουμε στην, στον ορισμό της αλληλείας μικρής κλίμακος. Αλλά λειτουργούν αυτοί οι στόλοι σε περιοχές που είναι σε ευαίσθητες και όπου πρέπει να υπάρξει προτιμησιακή εκμετάλλευση των πόρων και γι' αυτό χρειάζεται η επέκταση στο διάστημα 100 με 200 μίλια γιατί αν θέλουμε να μειώσουμε την πίεση στους αλληλευτικούς πόρους, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς που ιστορικά έχουν την πιο στενή σύνδεση με αυτούς τους πόρους να αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Και όχι απλώς να πούμε ότι οι στόλοι που είναι πιο ανταγωνιστικοί από οικονομική έποψη θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα αλωνίζουν εκεί. Αυτή είναι η λογική λοιπόν αυτή τη πρόταση. Άμα θέλουμε να υπάρχει ελευθερία πρόσβαση, όπω λέει και η κυρία Φράγα, αν η ελευθερία πρόσβασης είναι η βασική αρχή. Παράλληλα όμως θα πρέπει να έχουμε και ρυθμίσεις σε καταστάσεις όπου πρέπει να υπάρξει περιορισμός της πρόσβασης στους πόρους, ότι εκεί θα πρέπει στους περιορισμούς αυτούς να πριτανεύουν κριτηρία τα οποία δίνουν προτεραιότητα στην πρόσβαση αυτή στις αλλιευτικές κοινότητες που ιστορικά αλλιεύουν εκεί. Νομίζω ότι αυτό είναι πρέπον και ορθό και μέσα στο πλαίσιο αυτό έχω κάνει την πρόταση για τη διεύνηση της περιοχής ε, αποκλειστικής αλίας στα 200 μίλια. Γιατί είναι και ένας τρόπος με τον οποίο μειώνεται η πίεση στους αλληλευτικούς πόρους, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγκύτητα και ώστε το κέρδος από αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ευμάρεια των τοπικών αλλιευτικών κοινοτήτων. Θέλω λοιπόν να εξασφαλίσω αυτήν την ε, διατήρηση της ε, αποκλειστικής περιφέρειας για τις ε, υπερπεριφερειακές περιοχές ή τη διεύρυνσή της βάσει των ορίων της υφαλοκρηπίδας στις περιοχές αυτές αυτό το οποίο είπε η κυρία Μιράντα και ο κύριος Σάντσες Πεσέδο για τις δραστηριότητες παραδοσιακής ε, ηχθειοκαλλιάρκειας παρά το γεγονός ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί εδώ γιατί το αντικείμενο της έκθεσης ήταν η αλία εγώ πιστεύω ότι και πάλι για λόγους εγκύτητος θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια μνήμα για τα θέματα αυτά και ελπίζω ότι στις τροπολογίες σας θα μπορέσετε να συμπληρώσετε την έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να είναι γενικής αποδοχής και να είναι πλήρης η έκθεση. Και ένα τελευταίο θέμα που έθεσε η κυρία Λόβιν για την έννοια της ανανέωσης. Η ανανέωση αυτό είναι. Έχουμε καταστάσεις στις οποίες ορισμένα τμήματα της μικρής κλίμακος και αλλιευτικής ε, βιοτεχνικής αλίας γίνεται από σκάφη 20-30 ετών. Δεν τίθεται μονάχα ένα θέμα ασφάλειας για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στα πλοία αυτά, αλλά και θέματα αηφορίας για το περιβάλλον είναι αναποδοτικά σε σχέση με τη χρήση του καυσίμου τα πλοία αυτά και απλώς η πρόταση είναι να υπάρξει μια ανανέωση αυτού του στόλου που είναι πεπαλαιωμένος. Δεν μπορούμε να πούμε να πάρουμε αποφάσεις μηχανιστικές και τυφλές να πούμε ότι δεν θα υπάρξει ανανέωση του στόλου και ας πάνε να πνιγούν αυτοί μετά σαν πιο καραβάτους, θα πρέπει να κατανοήσουμε και ποια είναι η σημασία να έχουμε κοινωνική και περιβαλλοντική αηφορία μέσω μιας ανανέωσης η οποία θα λάβει υπόψη αυτή την πτυχή. Όχι να αυξήσουμε την αλληλευτική ικανότητα, αλλά να διατηρήσουμε την ανανέωση και να εξασφαλίσουμε τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα αηφορίας του περιβάλλοντος Όχι λοιπόν να πούμε ότι δεν είναι πια βιώσιμη αυτή η στόλη και θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Να δώσουμε μια δυνατότητα εξυγχρονισμού. Και σα τονίζω λοιπόν τα θέματα τη ασφάλεια και τη προστασία του περιβάλλοντο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέιρα. Σα υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 7η Μαΐου. 7 Μαΐου το μεσημέρι. Τα είπα αυτά προηγουμένως. Θα έχουμε πρόβλημα ε, επειδή θα υπάρξει ο χρόνος μετάφραση των ο, τροπολογιών πριν από τις 30-31 Μαΐου θα, δεν μπορέσουμε να συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε τον Ιούνιο. Αρχόμαστε <clears throat> στο σημείο 8, εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Λοιπόν, είπαμε θα είναι 8 ε, Μαΐου η προθεσμία, το μεσημέρι πάντα. Έχουμε εδώ πέρα μια έκθεση πρωτοβουλία σε σχέση με την εξωτερική διάσταση της αλληλευτικής ε, πολιτικής επί τη βάση μιας ε, πρότασης της Κομισιόν και αποφασίσαμε στην προηγούμενη μας συνεδρίαση να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων πριν από την υποβολή τροπολογιών σε σχέση με το θέμα αυτό και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούρη. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα αυτή να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων έχοντας λίγο περισσότερο χρόνο πλέον για την έκθεση αυτή. Σας έκανα μια πρώτη εισαγωγή στην προηγούμενη μας συνεδρίαση. Ουσιαστικά η έκθεση αυτή μιλάει από μόνη της. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που δραστηριοποιείται στην Αλία εκτός υδάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθεί και εκεί τις ίδιες προϋποθέσεις και τέτοια κριτήρια διαφάνειας, βιωσιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος με αυτά τα οποία ισχύουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ε, δυνατότητα αύξησης της ερευτικής ικανότητας και καθώς επίσης, έχουμε επίσης και κάποιες προτάσεις για την συμπερίληψη διμερών συμφωνιών. Προσδέπω λοιπόν συζήτηση που θα γίνει με τους συναδέλφους και στις ε, τροπολογίες που ενδεχομένω να καταθέσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στίβενσον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω την Ιζαμπέλα για την εξαιρετική αυτή εργασία που έχει κάνει, τις πολλές προσπάθειες που κατέβαλε. Είναι πολύ καλή έκθεση αυτή και πολύ απαραίτητη δεδομένου των συνθήκων. Όντως κάναμε συζήτηση στο παρελθόν. Ένα σημείο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι το ότι αναφέρεσαι στις απορρίψεις σε ορισμένα δηλαδή είδη τα οποία αλλιεύονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να προβλέπεται η ίδια απαγόρευση απόρριψη σαν αυτή που ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένων τώρα των προβλημάτων που έχουμε, προσπαθώντας να εξορολογήσουμε την απαγόρευση αυτή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή την απαγόρευση εκτός υδάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν επιβάλλουμε κάποιους πολλούς περιοριστικούς κανονισμούς στους δικούς μας τους στόλους, θα ήταν ιδιαίτερα άδικο αν όλοι οι υπόλοιποι που αλλιεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να κάνουν εκφόρτος, συγγνώμη, απόρριψη κάθε φορά που το επιθυμούν, ενώ για τους δικούς μας τους στόλους θα υπάρχει μια απαγόρευση. Θα βάλεις κάποιες κάμερες κλειστού κυκλώματος, θα υπάρχει ένα άλλο σύστημα παρακολούθησης. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Ο Σας ευχαριστώ, κύριε. Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, κριτήρια βιώσιμης αλίας και πρότυπα βιώσιμης αλίας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε ότι ο δικός μας ο ελευτικός στόλος θα είναι ανταγωνιστικός, ιδίως απέναντι στις λιγότερο υπεύθυνε χώρες. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την ανταγωνιστικότητα των δικού μας του στόλου με τα πρότυπα τα οποία ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όταν οι στόλοι βέβαια αυτοί δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν αβάσιμο όμως να λέμε ότι ε, ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μια προνομιακή σχέση όσον αφορά οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες σε βάρος των οικονομιών τρίτων χωρών ή σε βάρος αλληλευτικών κοινοτήτων τρίτων χωρών. Σε πολλές περιπτώσεις το σύνολο των αποθεμάτων παλιεύονται από τους στόλους αυτούς ουσιαστικά διοχητεύονται στην τοπική αγορά πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, οι πολίτες των χωρών αυτών έχουν πρόσβαση σε πιο φθηνά τρόφιμα. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει στην Δυτική Αφρική. Οι πόροι αυτοί δεν θα λιεύονταν ουσιαστικά αν δεν υπήρχαν ε, οι ε, κοινοτικοί στόλοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πράξουν κάτι τέτοιο. Η ελευτική μας λοιπόν πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη διαφόρων επαγγελματικών κλάδων σε τρίτες χώρες. Δεν θα πρέπει να κυνηγάμε απλώς το κέρδος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα κίνητρα στις τρίτες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν τα πρότυπά τους και την τεχνολογική ποιότητα των στόλων τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα πάρουμε από Ινστιτούτα όπως το FIO. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένου κανονισμούς. Υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κανονισμοί που θα κάναν τελικά τους δικούς μας τους τόλους λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με άλλους. και ξέρετε ότι θα μπορούσαν να βρεθούν διάφορε λύσει σε αυτό, μπορεί να οδηγηθούμε στο εξή φαινόμενο: να έχουμε κοινοτικού στόλου οι οποίοι θα φέρουν ξένη σημαία, σημαία τρίτη χώρα δηλαδή. Θα προετοιμάσω κάποιε τροπολογίες σε σχέση με τα αισθήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλέντσα. Ο κύριος Μιλάνα. Πάρα πολύ σύντομα. η εξωτερική διάσταση της ε, αλίας, δεν είναι μονάχα η οργάνωση της αλίας σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Το να εξασφαλίσουμε ότι η αλληλευτική μας πολιτική θα έχει επιτυχία και στην Ευρώπη και εκτός της Ευρώπης, αυτό απαιτεί μια σχέση με τον εξωτερικό χώρο που θα βελτιώσει τη συνολική κατάσταση και φυσικά θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αλληλευτικές συμφωνίες προβλέπουν ακριβώς την αλληλεία, την χρησιμοποίηση πόρων σε περιοχές που υπάρχουν ψάρια και όπου οι τοπικές αλληλευτικές ε, ικανότητες δεν είναι επαρκείς. Και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και η τοπική αλία και επίσης να δημιουργήσουμε μια αλλιευτική δραστηριότητα που βοηθάει τους Ευρωπαίους αλλιείς. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα αν η εξωτερική διάσταση της αλλίας, της ευρωπαϊκής αλλίας, δεν θα πρέπει να προβλέπει να υπάρχουν και αλλιευτικές συμφωνίες οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν την ικανότητα, τη δυνατότητα αλλιεύσης για ευρωπαϊκά σκάφη. Αναφέρομαι κυρίως στην ε, Μεσόγειο όπου μια συμφωνία θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχουμε τους ίδιους κανόνες αλίευσης και για τους ε, Ευρωπαίους αλίες και για τους μη Ευρωπαίους. Επίσης έχουμε την ε, Βουλγαρία, τους Βούλγαρους αλίες που αλίευουν στη Μαύρη Θάλασσα αλλά βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση με τους Τούρκους και Ρώσους αλίες που αλλιεύουν εκεί. Επίσης οι Ιταλοί και οι Ισπανοί βρισκόνται σε σύγκρουση με τους, με τους ε, Αλιερινούς ή τους ε, ε οι Έλληνες και οι Κύπροι με τη Βόρεια Αφρική κτλ. Με αυτές τις χώρες ε, έχουμε σχέδια και, και εξωτερική πολιτική. Άρα λοιπόν η μεταρρύθμιση της κοινή αρλευτικής πολιτικής μπορεί να λειτουργήσει έτσι ώστε οι συμφωνίες και οι πόροι που δίνονται σε αυτές τις συμφωνίες να είναι συμφωνίες που να μας επιτρέψουν να εφαρμόζουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για αυτές τις χώρες, για να σεβαστούν τους ίδιους κανόνες. Αυτό θα πει η οικοδόμηση πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για τις βόρειες θάλασσες, κάποιες από τις βόρειες θάλασσες. <coughs> όπου υπάρχουν όμορες χώρες. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να τεθεί αυτό το πρόβλημα σε αυτό το έγγραφο για να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε μία περίοδο που η εξωτερική πολιτική να μην είναι μόνο οργάνωση για την αλληλεία ορισμένων τόνων ψαριών σε μια θάλασσα που δεν είναι η ευρωπαϊκή. Αυτό δεν αποκαλείται εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι πάμε να, πάρουμε, να αγοράσουμε μερικά ψάρια γιατί τα δικά μας τελείωσαν. Ενώ το να πούμε εξωτερική πολιτική σημαίνει το, ε, να ε, οδηγηθούμε στο να υπάρξει μια ανάπτυξη θετική σε κάποιες θάλασσες, εξαλείφοντας τις συγκρούσεις και κυρίως έτσι ώστε οι πράξεις, οι δράσεις των πολιτικών μας να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Να κλείσω με ένα μικρό παράδειγμα, πολύ περιθωριακό σε σχέση με το ευρωπαϊκό βάρος, δηλαδή καλύπτει το 2%. Υπάρχει η σχεδόν κλειστή θάλασσα η Αδριατική στην Μεσόγειο. Από αυτήν βρέχονται η Σλοβενία και η Ιταλία που είναι κοινοτικέ χώρες, μια χώρα που είναι ένταξη, η Κροατία, και έπειτα το Μαυροβούνιο και η Αλβανία που βρέχονται από την ίδια θάλασσα. Σε αυτή τη θάλασσα σήμερα, σήμερα, ακόμα και σήμερα, η Σλοβενία και η Ιταλία αλλιεύουν στα ίδια νερά, όπου αλλιεύουν και οι Κροάτες. Οι Σλοβαίνοι και οι Ιταλοί σέβονται ή οφείλουν να σέβονται κάποιους κανόνες. Οι Κροάτες, οι Μαυροβούνοι και οι Αλβανοί όχι. Το αποτέλεσμα είναι ένα αριστούργημα. Και ποιο είναι αυτό το αριστούργημα? κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ανασύσταση των αποθεμάτων κτλ. Όλα αυτά ε, είναι μάταια. Και με τη ζημιά για την Ιταλική αλληλεία, Δηλαδή, οι αλληλεί μας δεν μπορούν να ψαρεύουν, οι άλλοι ψαρεύουν με διαφορετικούς κανόνες και αυτά τα προϊόντα έρχονται στη δικιά μα Ιταλική αγορά και ανταγωνίζονται τα ψάρια τα οποία έχουν αλληλευθεί με τον νόμο. Αυτή η κατάσταση ισχύει στην Αδριατική, στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, το Ανατολικό, στο κανάλι της Σικελίας. Και πρέπει να αλλάξει. Εμείς σήμερα αφήνουμε σε έναν, έναν γενικό ρόλο στις ε, διεθνείς συμβάσεις που είναι αυτοί οι σοφοί που συζητούν και που συχνά δεν σφίγγουν τα λουριά. Ε, και καθορίζουν αυτή την πολιτική. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο των αλληλευτικών συμφωνιών όπου η συμφωνία θα μιλά για τρόπο και όχι μόνο για αλίευμα. Παρακαλώ περιοριστείτε περιοριστεί τελικά στον χρόνο. Κύριος έχει το λόγο. Όταν μιλάμε για συμφωνίες βιώσιμης αλίας, σκέφτηκα το πρόγραμμα στη Βρετανική τηλεόραση, το Yes Minister, όταν θέλει κάποιος ε, ένας υπουργός να κάνει μια νομοθεσία που κάνει τα πράγματα πιο μυστικά, πρέπει να περιγράψει προς το κοινό αυτή την νομοθεσία ως αυτή που οδηγεί στη διαφάνεια. Γιατί ο κόσμος κοιτάζει τους τίτλους και όχι το περιεχόμενο. Λοιπόν, δεν θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό στην έννοια της αηφόρου αλίας. Κοίταζα τις τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος <clears throat> για το άρθρο που έχει να κάνει με τις ε, συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα στην Αλία. Τρία σημεία. Καταρχήν υπάρχει μια θέληση να λέμε ότι τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, αλλιεύουν σε αυτά τα νερά θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια όπω και στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αλλά πόσο πρακτικό χαρακτήρα έχει αυτό, σε ποιο βαθμό μπορεί να εξασφαλιστεί για τις απορρίψεις επίσης και για την υποχρέωση να εκφορτώνεται όλα τα ψάρια. Οι τροπολογίες αυτές παίρνουν την εξή γραμμή, λένε τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εκφορτώνουν σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα ψάρια τους ή σε άλλα λιμάνια που έχουν ειδική πιστοποίηση για να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι λογικό ή αν στέκεται ή αν είναι σε ένα φαντασιακό κόσμο όλα αυτά. Και τέλος <clears throat> το θέμα των σημαίων ευκαιρίας που αναφέρατε. Βλέπω να λένε τα μέλη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείε που έχουν βάσει στο Βερολίνο με σημαία Βενεζουέλα, παραδείγματο χάρη. Με πλοία που έχουν σημαία Βενεζουέλα. Και θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Και να βρούμε μια διατύπωση που να το εμποδίσει. Αλλά μου λέει η Κομισιόν. Μα Υπάρχει διεθνή νομοθεσία για τα θέματα αυτά και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτω τίποτα. Είναι έτσι. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιράντα. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την Ισαβέλα, ιδίω για αυτά που είπε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας για την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα κέρδος και για τον ευρωπαϊκό αλλιευτικό τομέα, αλλά και για να υπάρξει και μια ανάπτυξη της αλληλεκτικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές όπου πηγαίνουν τα πλοία μας. Η υποστήριξη σε προδιαγραφές αηφορίας επίσης, <clears throat> αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μεταξύ κρατών που εποφελούνται από αλληλευτικές συμφωνίες υπάρχουν συζητήσεις σε σχέση με την εγγύηση ότι είναι δίκαιες και αηφόρες αυτές οι συμφωνίες. Παραδείγματο χάρη για τη Μαυριτανία. Υπάρχουν ε, και στόλοι από άλλα κράτη-μέλη πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αλλιεύουν εκεί. Επομένως, στην εξωτερική διάσταση της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής υπάρχει αυτή η συμφωνία με τη Μαυριτανία που θα ε, περατωθεί τον Ιούνιο αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Υπότιτλοι θα τελειώνει τον Ιούνιο επιμένω <clears throat> στην ιδέα της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και στην αηφορία σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν 24 πλοία που αλλιεύουν κεφαλόποδα από την Ισπανία που δεν έχουν άλλο τρόπο αλλίες. Θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά τις διαπραγμάτευσεις εξωτερικής διάστασης αλλιευτικής πολιτικής. Πού μπορεί να υπάρξει τώρα κάποια διέξοδος όταν διακόπτονται συμφωνίες και όταν πάβουν να ισχύουν συμφωνίες, τι κάνουν αυτοί οι στόλοι που δεν έχουν εναλλακτικέ λύσεις, παραδείγματος χάρη ο στόλος που αλλιεύει στη Μαυριτανία, θα πρέπει και εδώ να βρεθούν κάποιες λύσεις κοινωνικής βιωσιμότητας όταν δεν υπάρχουν συμφωνίες ή όταν δεν ευδοκιμούν οι συμφωνίες. Τονίζω λοιπόν την αηφορία των πόρων, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική αηφορία. Ε, η κυρία Ροτόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Να προσθέσω κάτι θα ήθελα σε σχέση με αυτά που είπε ο Γκουίντο Μιλάνα. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Λέβεν, μάλλον κυρία Λόβεν, να πω καταρχάς ότι η εκθεσή σας είναι πολύ καλή. Όσον αφορά τώρα τα προβλήματα τα οποία έχουμε με τρίτες χώρες, αυτά τα σημεία αντιπαράθεσης, θα βρούμε κάποια λύση για αυτά τα προβλήματα, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια λύση, σε μια μελλοντική συμφωνία. Όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα, η ρήτρα αυτή αποκλειστικότητας αποτελεί τμήμα της απόφασης πλαίσιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι και απουσία πρωτοκόλλου θα εφαρμοστεί. Αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας, τότε οι πλειοκτήτες θα πρέπει να μπορούν να συνάπτουν μια συμφωνία με εκπροσώπους της τρίτης χώρας. Όσον αφορά το, τη ρήτρα υπαριθμών 15, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, σε σχέση δηλαδή με τις χώρες και τα μέρη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Και τέλος, η στόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά εξάγουν τα υψηλά μας πρότυπα σε τρίτες χώρες. Το ερώτημά μου λοιπόν το ακόλουθο. Οι τρίτες χώρες με τη σειρά τους θα συμμορφωθούν με τα υψηλά αυτά πρότυπα. Ή θα προσπαθήσουν τελικά να, βρουν λύσεις κάπου αλλού. Ο κύριος Σάντσες Περσέδο. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φιλοδοξήσει να είναι παγκόσμιος παίκτη στην αλληλευτική πολιτική και γι' αυτό <clears throat> θα πρέπει η Αλία να μπει και μέσα στην εξωτερική ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής και γι' αυτό, αυτό για πολλούς λόγους. Καταρχήν πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια ευθύνη σε σχέση με την προστασία της θάλασσας και των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και αυτό φυσικά ε, σημαίνει πρέπει να έχουμε ένα ρόλο σε διεθνείς οργανισμούς που διέπουν τα θέματα αλίας. Δεύτερον, οι συμφωνίες μας σε αλλιευτικό επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία στον αριθμό τους και όχι μια μείωση των συμφωνίων αυτών. Όχι μόνο να ανανεώσουμε αυτές τις συμφωνίες που έχουμε, αλλά να έχουμε περισσότερες συμφωνίες, να εδραιώσουμε την παγκόσμια μας αλληλευτική δραστηριότητα και να γίνει ένα κομμάτι της ε, πολιτικής μας ανάπτυξης και συνεργασίας η πολιτική αλίας. Ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 είναι η παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων και δεν μπορούμε εδώ να παραγνωρίσουμε την αλία που είναι μία από τις δραστηριότητες οι οποίες αποκτούν τον πιο διεθνοποιημένο χαρακτήρα. <clears throat> Αν θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο θα ισχύουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τους εταίρους μας, δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε ένα επίπεδο ιδιωτικοποίηση της αλίας. Θα πρέπει να υπάρξει μια δημόσια δράση, μια δημόσια ατζέντα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και όχι απλώς να ιδιωτικοποιήσουμε πλήρως την αλία. Δεύτερον, στην εξωτερική διάσταση, μια βασική πτυχή είναι οι εισαγωγέ αλληλευτικών προϊόντων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο για του καταναλωτέ μα, αλλά και για την αλυσίδα μεταποίησης αλληλευτικών προϊόντων. Εκεί θα πρέπει να επιλύσουμε λοιπόν όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί θα πρέπει η αλία να συμβάλλει στην τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς, αλλά και στη λογική λειτουργία της μεταποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα ένα θέμα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τις στρεβλώσεις στην εσωτερική μας αγορά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στην εξωτερική διάσταση την ανάγκη της αηφορίας και της ισότητος συνθήκων ώστε να μην υπάρχουν συστήματα αθέμητης, ε, αθέμητου ανταγωνισμού να μπορούν να είναι τέτοιες οι συνθήκες ανταγωνισμού που προέρχονται από τις συμφωνίες που να μην θέτουν σε μειονεκτική θέση τις ε, εταιρείες μας. Και αυτά είναι λοιπόν ζητήματα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ο κύριος Σαλαβράκος. Ε, πολύ λίγα θα πω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συγχαίρω την ε, κυρία Λέβεν για την ε, έκθεσή της. Είναι εξαιρετική. Ε, μελετώντας τι μου δημιουργήθηκε μελετώντας και την έκθεση του κύριου Φερέιρα ε, βλέπω ότι ίσως θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην άποψη του τι είναι ε, εξωτερικός χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Μεσόγειος, όπως είναι ο Εύξηνος Πόντος, η περιοχή του Εύξηνου Πόντου που έχει συμφέρον η Βουλγαρία και η Ρουμανία και να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας ίσως κανόνες το βάζω σαν προβληματισμό ε, ΑΟΣ, αντίστοιχες με την ΑΟΣ την αυτόνομη οικονομική ζώνη ούτως ώστε να δούμε οι συνθήκες ε, συνυπάρξεως με τα κράτη είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα γίνουν ευχερέστερα. Ε, σέβομαι όλες τις απόψεις που διατυπώνονται εδώ πέρα ως προς την ουσία του θέματος αλλά ε, ο προβληματισμός μου είναι γεωγραφικός και κατ' επέκταση της εκθέσεως. Ίσως θα πρέπει να ορίσουμε τις αυτόματες αλλιευτικές ζώνες, τις αυτόνομες αλλιευτικές ζώνες κατά τρόπο πιο καθαρό. Αυτά ήθελα να πω και να συγχαρώ και πάλι τη φίλη μας Σαβέλ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Η κυρία Γκαρτία Ιέρο. Πάρα πολύ σύντομα πρόεδρε. Για να συγχαρώ να συγχαρώ την ε, επικεφαλή στη γραμματεία που είναι γυναίκα και δεύτερον για να αναφέρω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Μιλάνα αλλά βλέπω να υπάρχει και μια σχιζοφρένεια όπου ανάλογα με την έκθεση λέμε διαφορετικά πράγματα. Έχουμε τρία βασικά έγγραφα σε σχέση με τα οποία έχουμε την συναπόφαση και έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση ως κοινοβουλευτική και οι τροπολογίες που τίθενται είναι αντιφατικές. Από την ίδια πλευρά θέλουμε να ψαρεύουμε πολύ οι εφοπλιστές μας να έχουν πολύ καλές συνθήκες αλίευσης και από την άλλη πλευρά θέλουμε να διατηρήσουμε όλες αυτές τις βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την βιωσιμότητα του θαλάσσιου χώρου κτλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές και περιοχές οι οποίες ε, καλύπτονται από πολλές χώρες, κάποιες από τις οποίες δεν είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε μια συνεκτικότητα στην θέση μας. Δεν μπορούμε να θέτουμε στον εαυτό μας περισσότερα προσκόμματα από ό,τι μας θέτει το διεθνές δίκαιο στο οποίο υποκείμεθα. Αν θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι και στις τρίτες συμφωνίες με τρίτες χώρες ότι έχουμε ένα το πλαίσιο που έχουμε μάλλον συμφωνήσει με τρίτες χώρες δεν μας επιτρέπει να τους επιβάλλουμε τα δικά μας πρότυπα. Θα πρέπει να συζητήσουμε σε λίγο τις ε, τροπολογίες για την ε, ε, ελεύθερη οργάνωση της αγοράς. Δεν μπορούμε όμως να συζητάμε θέματα της αλίας ανεξάρτητα από αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που συζητά εν γέρι το Κοινοβούλιο. Ο κ. Μπέρκ από την Κομισιόν. Bonjour. Non, Σας ευχαριστώ πολύ. που μου δώσετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση βάσει μιας εξαιρετικής έκθεσης από την κυρία Λεβίν. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά σημεία κατά την άποψή μου όσον αφορά την μεταρρύθμιση των συμφωνιών αλίας και της εξωτερικής διάστασης αλίας είναι καταρχάς πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον ρυθμιστικό χαρακτήρα αυτών των ελευτικών συμφωνιών. Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο πλαίσιο δραστηριότητας θα μπορούσαμε να είχαμε όσον αφορά τους κοινοτικούς στόλους στο εξωτερικό. Το ρυθμιστικό λοιπόν αυτό χαρακτήρα τον υπογραμμίζει η έκθεση και θα πρέπει βέβαια να τον βελτιώσουμε, να τον μεταρρυθμίσουμε, διατηρώντας όμως το πλαίσιο αυτό προκειμένου να έχουμε συμφωνίες βιώσιμης αλίας. Θέλουμε στα διεθνή ύδατα και στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, προκειμένου οι συμφωνίες αυτές να είναι πραγματικά βιώσιμες. Να λαμβάνουν υπόψη τους τους ελευτικούς πόρους, οι οποίοι δέχονται όλο και υψηλότερε πιέσεις. Στόχος μας είναι να δυναμώσουμε τη διακυβέρνηση και να ενισχύσουμε την συνέπεια με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εμπορική πολιτική για παράδειγμα, το αναφέρατε αυτό, με την πολιτική ανάπτυξης κτλ. Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε στις τρίτες χώρες την επίπτωση που έχουν αυτές οι συμφωνίες. Και συγκεκριμένα φέρομαι στην προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από τις συμφωνίες αυτές οι χώρες εταίροι μας. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να επενθυμίσουμε ότι ε, ο εξωτερικός αυτός στόλος δεν βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τον τοπικό στόλο με τον βιοτεχνικό, αν θέλετε, στόλο, το στόλο βιοτεχνικής αλίας των τρίτων αυτών χωρών. Συχνά προωθείται η άποψη αυτή. Βρισκόμαστε όμως σε ανταγωνισμό με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία ή και άλλες χώρες, οι οποίες αλλιεύουν σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων χωρών, έχοντας χαμηλότερο επίπεδο διαφάνειας και παραθέτοντας χαμηλότερε εγγυήσει από αυτέ που εμεί απαιτούμε στα πλαίσια των ελευτικών μα συμφωνιών. Πρέπει λοιπόν να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο να καταφέρουμε να αυξήσουμε την επιστημονική διάσταση των ε, συμφωνιών αυτών και να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία και με την κερδοφορία των ε, συμφωνιών αυτών. Ένα ιδιαίτερο ερώτημα ακούστηκε. Αν θα μπορούσαμε να έχαμε αληφτικές συμφωνίες χωρίς ε, δικαιώματα πρόσβασης στους ε, πόρους. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε όμως κάπως περισσότερο, θα χρειαστεί να τη μελετήσουμε από κοινού. Όσον αφορά τώρα το κείμενο της έκθεσης, το επαναλαμβάνω ότι η έκθεση Λεβίν είναι μια εξαιρετική έκθεση, ωστόσο έχουμε κάποιες ανησυχίες ή παρατηρήσεις για κάποια συγκεκριμένα σημεία. Καταρχάς η ρήτρα της αποκλειστικότητας. Αναφέρεται σε αυτήν η έκθεση και θεωρεί ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί η ρήτρα αποκλειστικότητας. Δεν ξέρουμε αν απαραίτητο κάτι τέτοιο Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ρήτρα αποκλειστικότητα, αλλά κάθε φορά που εφαρμόζεται, κάθε φορά που συμπεριλαμβάνεται σε μια συμφωνία και όχι στο πρωτόκολλο, καταλήγουμε σε καταστάσει μπλοκαρίσματο κάθε φορά που δεν ανανεώνεται το πρωτόκολλο για τη μία ή την άλλη περίπτωση, όπω συμβαίνει ήδη με κάποιε συμφωνίε μα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάθε φορά που λέμε ότι θέλουμε να δυναμώσουμε υπερβολικά αυτή τη ρήτρα αποκλειστικότητα. Τώρα, όσον αφορά την συμβολή των πλειοκτητών στο κόστος πρόσβασης και στο κόστος των συμφωνιών αυτών εν γέννη, Ας είμαστε και εδώ προσεκτικοί και ας έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και ας υπενθυμίσουμε ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει μια εξισορρόπηση των, της συμβολής των εφοπλιστών, των πλειοκτητών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δεν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα όπου το σύνολο του ποσού θα καταβάλλεται από τους πλειοκτήτες. Στην περίπτωση αυτή, οι συμφωνίες δεν θα είναι ελκυστικές για τις τρίτες χώρες που δεν θα έχουν το εγγυημένο αυτό εισόδημα το οποίο προέρχεται από την καταβολή που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προπολογισμού της. Market-based approach, προσέγγιση βάση της αγοράς. Ναι, αλλά με κάποιους περιορισμούς και εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αυτό και θα πρέπει οι πλειοκτήτες να καταβάλουν βέβαια φόρους, τέλη, κάθε φορά που αλλιεύουν σε τα τρίτων χωρών. Πέρα από την άδεια υπάρχουν και κάποια τέλη όσον αφορά την ναύλωση, όσον αφορά την παρουσία παρατηρητών και το καθεξής. Δηλαδή τέλη τα οποία προστίθενται στην πληρωμή της άδειας. Καταλαβαίνω επίση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να πετύχει μια διαφάνεια, καθώ επίση και μια παρακολούθηση των ε, συμφωνιών αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εξωτερικού παρατηρητέ. Αν όμω ε, για κάθε συμφωνία αυξάνουμε τις εκθέσεις σε αιτήσια βάση όπως προτείνεται, θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα που τελικά θα πνιγούμε από όλες αυτές τις αναφορές που θα μας καταφθάνουν ανα πάσα στιγμή. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να γίνεται μία έκθεση αξιολόγησης κάθε φορά που θέλουμε να ανανεώσουμε ένα πρωτόκολλο. Θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη παρακολούθηση στα πλαίσια των μεικτών επιτροπών. Και βέβαια οι μεικτές αυτές επιτροπές είναι ανοιχτέ και για σας και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται τώρα να προβλέψουμε τόσες πολλές επιπλέον εκθέσεις που άλλωστε δεν θα μπορούσαμε καν να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ήταν σε θέση να εξετάσει όλες αυτές τις εκθέσεις, όλες αυτές τις αναφορές για την υλοποίηση και εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα να κάνω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Λέβεν για να κλείσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τα ερωτήματά τους και για την υποστήριξη που μου έχουν δώσει. Να ξεκινήσω με αυτά που είπε η Κομισιόν. Δεν αληθεύει απόλυτα και σε κάποιες περιπτώσεις δεν αληθεύει καθόλου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταγωνίζεται με τους τοπικούς στόλους και απλώς ανταγωνίζεται άλλους διεθνείς στόλους. Υπάρχουν περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλιεύει τόνο παραδείγματος χάρη, τον οποίο ψαρεύουν και οι τοπικοί στόλοι, αλλά σε διαφορετικές περιοχές. Οι τοπικοί στόλοι σε παράκτια ύδατα και η Ευρωπαϊκή ή άλλη στόλοι σε πιο ανοιχτή θάλασσα. Για τη Μαυριτανία παραδείγματος χάρη τα χταπόδια αλλιεύονται και από τον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους τοπικούς ψαράδες. Τα θέματα της αποκλειστικότητος είναι σημαντικά. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Σάντσες Πρεσέρο, να πούμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τμήμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, αν θέλουμε να παροτρύνουμε την βιώσιμη αλία και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιδέα ότι ο φορολογούμενος θέλει να εμπλακεί σε όλα αυτά είναι να υποστηρίξουμε την βιώσιμη αλληλεία στις χώρες αυτές. Αν πληρώνουμε απλώς για την πρόσβαση ορισμένων πλοίων και κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτά που κάνουν οι στόλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το χώρο της συμφωνίας, αυτό δεν δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπευθυνότητα στα θέματα αυτά γινόμαστε ερεντίκολο των σκυλιών. Ακολουθούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά με τον τρόπο αυτό. Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια εξωτερική διάσταση θα πρέπει να τηρήσουμε και το πνεύμα και το γράμμα των συμφωνιών. Και θα ήθελα να ενισχύσω ακόμα περισσότερο αυτό το επιχείρημα γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν με άλλες σημείες σημαίες στο Κάμπο Βέρντε. Έχουμε πλοία τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά στα χαρτιά, γιατί δεν έχουν ευρωπαϊκή σημαία, αλλά στην πράξη είναι ευρωπαϊκά. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά αντίθετα πιο σφιχτοί. Και τώρα για τη συμβολή των εφοπλιστών. Να σας υπενθυμίσω ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια Μεγάλων Αποστάσεων είχαν συμφωνήσει να δίνουν ένα δίκαιο τίμημα οι εφοπλιστές για την πρόσβαση σε αυτά τα ύδατα. Και δεν θεωρώ ότι αν πληρώνανε περισσότερο θα είχαν λιγότερο ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτές τις συμφωνίες. Έχοντας συζητήσει με πολλούς εκπροσώπους του στόλου αυτού μεγάλων αποστάσεων, θεωρούν ότι είναι πολύ ελκυστικό να καλύπτονται από την νομική ασφάλεια μια συμφωνίας που εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς μπορεί να φύγονται από την ε, ανασφάλεια των συνδικών αυτών. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές στα θέματα αυτά. Ο στόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τόνο πληρώνει 35 ευρώ τον τόνο στον Νότιο Ειρηνικό θέλουν 5 ή 6 δολάρια την ημέρα. Δεν είναι λοιπόν τα 35 ευρώ για τον τόνο είναι ελάχιστο ποσοστό της πραγματικής αξίας των αλλιευμάτων. Στο όνομα λοιπόν της ισοδικίας για όλους τους στόλους σε παγκόσμιο επίπεδο, εμείς δεν θα πρέπει να επιδοτούμε τους επιχειρηματίες, θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο τίμημα πρόσβασης, γιατί και πριν από όλα αυτά τα πράγματα ήδη τους υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαπραγματεύεται εξ ονόματός τους, κάνει την αξιολόγηση και όλα αυτά τα πράγματα. Οι φορολογούμενοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο για να προωθήσουν μια βιώσιμη πολιτική εκμετάλλευση των θαλασσών. Και μόνο για αυτό το λόγο. Και όταν πρόκειται για τις ανησυχίες της Κομισιόν ότι θα έχουν τεράστιο χαρτοβασίλειο να αντιμετωπίσουν και αξιολογήσει. εγώ πραγματικά ενκπλήτωμαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρει πάρα πολλές αξιολογήσεις και βλέπουμε ότι δεν υπήρξαν μικτές επιτροπές συναντήσεις των μικρών επιτροπών αντίθετα από αυτά που λέγονται σε άλλες συμφωνίες. Παραδείγματος χάρη συμφωνία με τη Μοζαμβίκη. Στην αρχή δεν υπήρχαν καθόλου συναντήσεις των μεικτών επιτροπών και είδαμε στην αξιολόγηση που ακολούθησε ότι δεν υπήρξε καμία ε, βελτίωση στην εθνική αλία της Μοζαμβίκης, δεν υπήρξε η παραμικρή υποστήριξη στον αλληλευτικό τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αν θέλουμε να συνεχίσουμε τέτοιου είδου συμφωνίε, ενώ τι βαφτίζουμε ότι είναι αηφόρο, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχουν αξιολογήσει, θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα προτού πούμε ναι, ναι, εγκρίνοντα μια τέτοια συμφωνία στο μέλλον. Αυτό ισχύει και για το Συμβούλιο. Οι κοινοβουλευτικοί στα κράτη-μέλη. Και αυτοί θα πρέπει να έχουν ένα ρόλο σε όλα αυτά. Δεν ξέρουν τίποτα. Αν η κυβέρνηση στην Σουηδία πει ότι είναι καλή αυτή η συμφωνία, θα πει και το Κοινοβούλιο ναι, αλλά δεν έχουν δει την παραμικρή έκθεση αξιολόγηση για όλα αυτά τα θέματα. Συγγνώμη, μπερδεύαμε μερικές φορές. Λοιπόν, κανείς δεν έχει την πληροφόρηση για αυτά τα θέματα. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτή η δημοκρατική ε, διαφάνεια. Ίσως έπρεπε να μιλήσω σου ειδικά, αλλά όλα τα έγραφα είναι στα αγγλικά και είναι πιο εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ υπερβολικό αριθμό συναντήσεων των μεικτών επιτροπών, υπερβολικό αριθμό αξιολογήσεων, εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αποτελεσματικότητα να υπάρχει αηφορία. Αλλιώ δεν πρέπει ούτω ή άλλω να κάνουμε συμφωνίε αυτό το είδου. Για του συναδέλφου, για τα ερωτήματά του. Για τι απορρίψει. Υπήρξαν κάποια ερωτήματα για τι απορρίψει. Σε όλε σχεδόν τι συμφωνίε υπάρχουν προβλέψει για παρατηρητέ στα σκάφη. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξει κανείς τα θέματα συμμόρφωσης από ό,τι στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μου ανησυχία είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει σαν αποτέλεσμα ένα είδος dumping τιμών σε τοπικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ξέρω ότι οι γαριδάδες στη Γουινέα Μπισάου μπορούν να έχουν 80% παράπλευρα αλλιέματα. Αν τα πάει κανείς όμως αυτά στην τοπική αγορά, τι γίνονται οι τοπικοί ψαράδες. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το dumping των τιμών. Υπάρχει πάντα συζήτηση όμως για τις απορρίψεις ηχθείων. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να προωθήσουμε μια βιώσιμη μορφή αλίας, θα πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία και να μην επιτρέπουμε να μην επιβάλλουμε μια σειρά κανόνων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτι αντίθετο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μιλάνα, μας φαίνεται αυτές τις επαναστατικές σας ιδέες και πάλι. Αυτό το οποίο προτείνουμε και αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση που προκρίνεται εσείς να υπάρξει αποσύνθεση της πρόσβασης στην Αλία με την υποστήριξη στον αλληλευτικό τομέα. Αν έχετε πλήρη αποσύνδεση, μετά δεν χρειαζόσαστε να υπάρχει συμφωνία για πρόσβαση. Μπορείτε να έχετε μονάχα την τομεακή υποστήριξη. Ναι, δεν είναι τόσο παράλογο. Όλη η λογική πίσω από την αποσύνδεση είναι Παραδείγματο χάρη, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα σκάφη της οδηγεί σε υπερβολική αλεία, μεταφεύγουμε και παίρνουμε και την υποστήριξη στον αλλιευτικό τομέα μαζί μας. Και άμα είναι μια φτωχή χώρα, αυτό είναι ανήθικο. Έχουμε καθαρίσει τα ψάρια τους και μεταφεύγουμε κιόλα. Μια αποσύνδεση θα επέτρεπε να υπάρχει τομεακή υποστήριξη στην αλία χωρίς αλληλευτική δραστηριότητα. Αυτό θα ήταν απόλυτα δίκαιο και συνεκτικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχει βοήθεια κάτω από συνθήκες εξάρτησης, όπως ε, έχει συμβεί με όλες τις αλληλευτικές συμφωνίες μέχρι τώρα. Πώς θα βελτιώσουμε όμως τη σχέση με τις χώρες αυτές στη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, <clears throat> την Αδρία. Σημαντικά είναι αυτά τα ερωτήματα. και εξεπλάγει όταν υπήρξε αυτή η έκθεση της κυρίας Ρότοβα που τόνισε ότι δεν υπάρχει συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα. Μα εδώ είναι βασικό στοιχείο διαχείρισης αλληλευτικών πόρων. Θα πρέπει να συνεργάζεστε με τις χώρες που ψαρεύουν τα ίδια ψάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να δείξει μεγαλύτερη δραστηριότητα και ίσως εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Για τον κύριο Ντέιβις, για τις ε, βιώσιμες αλληλευτικές συμφωνίες. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα ή κάποιο γκαϊλέ για τις αλλαγές ονομάτων. Υπάρχει πρόταση κομισιόν να αλλάξουμε τα ονόματα. Ίσως ένας λόγος για να αλλάξουμε τα ονόματα, να υποστηρίξουμε μια αλλαγή ονομάτων, είναι γιατί λέμε ναι, τώρα έχουμε μια νέα γενιά συμφωνιών Οπότε μπορείτε να κάνετε μία διάκριση από τις παλιές αλλιευτικές συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα. Αν μας πείραζε η λέξη βιώσιμη, αν νομίζαμε ότι θα μας κοροϊδέψουν, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα μας κοροϊδέψουν για την έννοια της εταιρική σχέσης, γιατί δεν είναι εταιρική σχέση όπως ξέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να εξασφαλίσουμε ότι οι αλληλευτικές συμφωνίες θα είναι βιώσιμες. Μα γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις εκθέσεις ε, αξιολόγησης της συνεδριάσεις των μεικτών επιτροπών, τους ελέγχου και τους παρατηρητές στα σκάφη, που δεν έχουν γίνει πραγματικότητα στο παρελθόν, πολλές φορές. Για τις σημαίες ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε βέβαια τις σημαίες ευκαιρίες και αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, γιατί πάντα το κράτος σημαίας έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων, αλλά όταν πρόκειται για τελικούς ιδιοκτήτες που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και τα κατημέρια μελη θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά είναι και θέμα πολιτικής θέλησης να προσπαθήσει κανείς να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. και σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Παραδείγματο χάρη στην Σιέρα Λεόνε είχαν ανοιχτό νεολόγιο που θα μπορούσε ο καθένα να πάει να εγγραφεί στην σημαία τη Σιέρα Λεόνε. Και όταν ο Υπουργό Αλία στη Σιέρα Λεόνε ήρθε, τον πλησίασε μία μήκυο και του εξήγησε τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, είπανε ωραία, κλείνουμε το νεολόγιο. Δεν ήταν τόσα πολλά λεφτά που έβγαζε η Σιέρα Λεόνε, ήταν απλώς ότι δεν ήταν κάτι το οποίο είχε μεγάλη σημασία σε πολιτικό επίπεδο για αυτούς. Τέτοια προβλήματα λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ναι, ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου. Λέει ο πρόεδρος. Πηγαίναμε πολύ καλά. Αλλά στο προηγούμενο και το προ-προηγούμενο σημείο έχουμε έχουμε μακρηγορήσει. Μας μένει ένα σημείο ακόμα στην ημέρησια διάταξη που είναι η έκθεση του κυρίου Μπεσέτ. Για να τελειώσουμε τώρα σε 6.30 βέβαια δεν προφταίνουμε. Εγώ προτείνω να θέσουμε το σημείο του κυρίου Μπέσετ αύριο, οπότε θα έχουμε και το 9 του κυρίου Ρωμέβα και το 9α, εάν συμφωνεί ο κύριος Μπέσετ. Οπότε μέχρι τις 6.30 μπορεί η κυρία Λέβιν να απαντήσει προς πάντα ενδιαφερόμενα. Κύριε Μπέσετ, εντάξει. Ναι, ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Έχετε ακόμα 7-8 λεπτά για να κλείσετε, κυρία Λέβεν. Απαντούσα σε όλους τους βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέσετ. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είδα το ρολόι. Συγγνώμη, Ζαν Πολ. Δεν ε, ήθελα να μιλήσω τόση ώρα. Σάντσες Πεσέντα, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παγκόσμιος παίκτης, ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες συμφωνίες. Εγώ συμφωνώ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίζει παγκόσμιο ρόλο, αλλά όχι περισσότερες συμφωνίες με κάθε κόστος, με κάθε τίμημα. Ήδη έχουμε πολύ ουσιαστικά προβλήματα με κάποιες από τις συμφωνίες που ήδη έχουμε κάνει και θα πρέπει να διορθώσουμε λίγο το σχέδιο τους πριν να προβούμε και σε νέε συμφωνίε. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να είναι αξιόπιστη, θα πρέπει να έχουμε κάτι που καλό να δείξουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως το έχουμε. Αλλά ελπίζω πως θα το έχουμε στο μέλλον. Κυρία Γκαρσία Χιέρο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε μόνο στι εθνικά συμπεφωνημένε αρχέ και να μην προχωρήσουμε άλλο, αλλά είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να πάμε προ τα πάνω και όχι προ τα κάτω. Να προχωρήσουμε δηλαδή όσο γίνεται για να προωθήσουμε τη βιώσιμη αλληλεία στι περιπτώσει που οι γείτονε δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω τελείωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λέβεν. 8 Μαΐου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες της έκθεσης αυτής. Αύριο στις 9 το πρωί με τη βοήθεια του Θεού θα ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό της Νορβηγίας για την αλληλεία και τα παράκτια θέματα. Σας παρακαλώ να έρθετε στις 9 για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εν και να μην καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο στην ίδια αίθουσα. Αύριο στις 9 και ευχαριστούμε τους διερμηνείς.